Guten Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Καλώς ορίσατε θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου. Έχετε τριμερήσια διάταξη, δεν ε, έχουν ζητηθεί αλλαγές εξ όσο γνωρίζω, ε, μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο. Χαιρετίζω τον παγκόσμιο τύπο. Έχουμε νέο μέλος, τον κύριο Κον, από τους ε, ε, ε, Σοσιαλδημοκράτε, συγγνώμη, χαιρόμαστε για κάθε ενίσχυση που έρχεται στην Επιτροπή μα. Ε, σημείο 2, στην ημερήσια διάταξη, ε, είναι οι γλώσσε που μπορείτε να βρείτε και στο Cont News που έχουμε. Στι 4 έχουμε ψηφοφορίε και σα παρακαλώ να ετοιμάσετε τις κάρτε σα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 13 Φεβρουαρίου και 27-28 η Φεβρουαρίου είναι στη διάθεσή σας και αν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν έχετε εκφράσει επιθυμία για αλλαγές ή αντιρρήσεις, ε, θεωρούνται εγκεκριμένα. Σημείο 4. Σχέση κόστους αποτελεσματικότητας του 7ου προγράμματος έρευνας. Συγγήτρες είναι η κυρία Διάμπα Χοβά και η κυρία Σέντερ. Δυστυχώς ε, ασθενή η κυρία Σέντερ Πρόσφατα ε, Θα μάθαμε περαστικά. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λαμπαχοβά και λόγω της ασθένειας της κυρίας Αγιαλασάνη μάλλον θα χρειαστεί παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών που θα είναι 3η-4η Απριλίου. Θα το δούμε αυτό μέχρι το τέλος της ε, συζήτησης. Ε, το λόγο έχει η Μαρτίνα Λαμπάχοβα. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που απουσιάζει η Νέσ και δεν μπορεί να είναι μαζί μου εδώ. Την αντικαθιστώ βέβαια, αλλά όπως βλέπετε και από το σχέδιο έκθεσης είναι κοινό πόνημα. Θα προσπαθήσω να κάνω μία σύντομη ε, παρουσίαση και να ακούσω κυρίως τα σχόλιά σας και να τα μεταφέρω και στην Ινέση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η συνεργασία μας επί του σχεδίου αυτού ε, έκθεσης. Ε, επικεντρωνόμαστε στην προστιθέμενη εξή και στην αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι, αυτή είναι και η στο συγκεκριμένου έκθεση και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι γενικώ ε, ήταν αποτελεσματικό το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και ελήφθησαν υπόψη οι προτάσει μα κατά τη διαχείριση αυτού του προγράμματο ε, την ευχαριστούμε ότι αφουγκράστηκε τον προβληματισμό μα. Ε, έχουμε 55 δις ε, προϋπολογισμό 3% των συνολικών δαπανών ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, το 25% της ανταγωνιστικής χρηματοδότησης ε, γενικώ. Και μάλιστα στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η ομάδα ψηλού επίπεδου το Δεκέμβριο του 2015. Θεώρησε και αυτή η ομάδα επιτυχές στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και επισήμανε ότι ενθαρρύνει την αριστεία σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο, προωθεί την πρωτοποριακή έρευνα μέσω του καινοτόμου ειδικού προγράμματος ιδέες του 7ου ε, προγράμματο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. διασφάλισε τη συμμετοχή τη βιομηχανία και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στρατηγικό τρόπο, πρόθεσε ένα τρόπο συνεργασία νέο και ένα πλαίσιο ανοιχτή καινοτομία και επίση δημιούργησε ολοκληρωμένα δίκτυα ικανών να ανταποκρίνονται σε θεματικέ προκλήσει. ενώ ταυτόχρονα έδωσε ενάψματα για την κινητικότητα των, κινητικ... των ερευνητών στην Ευρώπη ε, και δημιούργησε μια ανοιχτή αγορά των ε, ερευνητών και ανοιχτή αγορά εργασία. Επίση, πρόθεσε τι επενδύσει σε ευρωπαϊκέ ερευνητικέ υποδομέ και κατά την επταετή περίοδο ε, ε, λειτουργία του προγράμματο, 130.000 περίπου ερευνητικέ προτάσει υποβλήθηκαν και επιλέχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν 25.000 έργα ύψη ποιότητα. Οι κύριοι αποδέκτε μεταξύ των 29.000 οργανισμών που συμμετείχαν στον 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ήταν πανεπιστήμια. Το 44% τη χρηματοδότηση το διεκδίκησαν τα πανεπιστήμια από το πρόγραμμα αυτό. Ενώ οι οργανισμοί έρευνα και τεχνολογία είναι σε δεύτερη θέση, 27%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 13%, 13% και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις 11%, 11 της χρηματοδότησης. Βέβαια, εντοπίσαμε και κάποιες στενοπούς που θα πρέπει να αρθούν χάρη του εξυγχρονισμού που προσφέρει το ορίζοντας 2020 και να θα εφαρμοστούν κατά την προετοιμασία του ένατου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Θέλουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα μεταξύ των προπολογισμών των υποπρογραμμάτων σημαντική αυτή η ανάγκη ενίσχυση τη ε, ευελιξία, κατά αποκοπή ποσά για τα έμεσο κόστο, μια νέα στρατηγική λογιστικού ελέγχου, αυτό το τονίζουμε και το επισημάναμε και στο σχέδιο έκθεση, ένα ενιαία δικτυακή πύλη συμμετοχή και κάποιε άλλε στάσει που προτείνουμε στο σχέδιο έκθεση. Επίση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το θέμα του Brexit, γιατί ξεκινάει η, ομάδα, η εβδομάδα Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταλήψει την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο από δημοσιονομική άποψη, αλλά και άποψη ε, μελλοντική συνεργασία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Γιατί είχαμε πολλέ μεικτέ ομάδε με συμμετοχή Βρετανών ερευνητών και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και μάλιστα οργανώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν 1,27 δις 2000, ε, από το 2013 και είναι 15% του 1,18 δις από τους διαγωνισμούς. Ε, ε, είναι πολύ μεγάλο το μερίδιο, μεγαλύτερο μερίδιο ε, χώρες μέλους μεμονωμένης από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον αυτής της συνεργασίας με το Μένο Βασίλειο, με ερευνητικές ομάδες που έχουν τη βάση του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι θα γίνει στο μέλλον με αυτή τη συνεργασία. Επίσης, ε, θέματα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, ε, θέμα χρηστής οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης για να υλοποιήσουμε τους στόχους πολιτικής. Σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης φυσικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αντικειμενικά ε, γιατί αυτή τη, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Ακόμη ε, και με μονομένα σχέδια μπορούν να προωθήσουν την έρευνα, ακόμη και αν αρχικά δεν θεωρούνται επιτυχημένα. Και αυτή είναι η πρόκληση για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, να βρούμε τα πραγματικά ωφέλη, τα πραγματικά επιτέγματα. Θα βάλω τελεία εδώ, γιατί με ενδιαφέρουν κυρίως τα σχόλια των συναδέλφων και περιμένουμε και τις τροπολογίες σας, τα σχόλιά σας για την έκθεση και θα ευχαριστήσω θερμά και την Ινές για την πολύ καρποφόρα συνεργασία που είχαμε και προσβλέπω και στην μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση για την έρευνα. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Την μελετούμε με πολύ ενδιαφέρον. Πολλά θετικά βλέπουμε. Κάποια χρειάζονται μια βελτίωση. Με πολύ μεγάλη σοβαρότητα βέβαια το μελετούμε. Μαζί σας έχουμε άλλη μια κρόαση σε κάνα δύο μήνες. Κρόαση που πιστεύω θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό του ένα του προγράμματος. Έχουμε καλές επιδόσεις προς την υλοποίηση του ορίζον 2020. Κοιτούμε τους στόχους πολιτικής, το πιο σημαντικό που έχουμε να επιτελέσουμε. Η αποτελεσματικότητα βέβαια και το κόστος, ο λόγος αποτελεσματικότητας προς το κόστος είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο αντικειμενικά να αποδειχθεί. Είναι χρήσιμα κάποια από τα στοιχεία της έκθεσης για τους υπολογισμούς αποτελεσματικότητας και κόστους. Προσπαθούμε να τα ενσωματώσουμε και στις αιτήσεις έκθεσης ε, παρακολούθησης, ώστε να είναι πιο ορατή για σας κάθε χρόνο πως προχωρεί το πρόγραμμα ε, αυτή η διάσταση, να μην αφήνουμε δηλαδή στο τελικό, στην τελική έκθεση να καταγράφεται μόνο. Για το Brexit ξέρετε ότι δεν έχω εντολή να επεκτείνουμε στο θέμα αυτό. Ξέρουμε βεβαίως όλοι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντικός εταίρος στο πρόγραμμα πλαίσιο. Όλοι μας στην Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και την Τεχνολογία ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η συμμετοχή του. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι Βρετανοί ερευνητέ το ίδιο επιθυμούν αλλά ασφαλώς αυτό θα κρυθεί από τις διαπραγματεύσει για τις οποίες δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να επεκταθώ. Ευχαριστούμε για την έκθεση και προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία μέσα σας και την πορεία προς το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα υπολογίσει ότι θα ακούσω πρώτα τι έχετε εσείς να πείτε γιατί είχαμε κάποια ζητήματα με το πρόγραμμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω πόσες διαδικασίες έχετε ενώπιον του δικαστηρίου, για ποια κράτη, ποιες διαδικασίες έχει αναλάβει η Όλαφ, ποιες έχει ολοκληρώσει, ποιες ακόμα είναι κρεμείς. Και θα ήθελα επίσης, γιατί αναφέρεται στην έκθεση ότι 95, ε, 59% των ε, ποσών που ε, ότι το 59% είναι αυτό το ποσοστό των ποσών που επαληθεύονται. Τα υπόλοιπα τι γίνονται. Για τα καταποκοπήν ποσά επίσης. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία πώς τα αντιμετωπίζετε και τι είδους συμπεράσματα αποκομίζετε για το μέλλον, για τα καταποκοπήν ποσά. Αυτά ξεκινώντας και δίνω το λόγο, εάν δεν θέλει άλλος συνάδελφος, στην κυρία Βουέπ. Okay. Um, Στον κύριο Κοιτάξτε, για τις ε, δίκες και τις υποθέσεις Όλαφ θα πρέπει να σας δώσω γραπτή απάντηση. Για την έρευνα και τεχνολογία λίγο πολύ έχω στοιχεία αλλά είναι και άλλες οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Επομένω καλύτερα να τα ε, καλύψω σε, ένα, σε μια γραπτή απάντηση. Το 59% λοιπόν ελέγχεται. Καλύπτονται από τις εκθέσεις των ελεγκτών. Ε, εάν όμως υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχουμε τρεις ε, διεκδικήσεις από ζημίωσης με έγκριση τότε συνήθω προβλήματα δεν υπάρχουν. Εάν μπορεί να γίνει μια διόρθωση, τότε προχωρούμε. Στο 59% έχουμε μια άμεση ή έμεση κάλυψη, λίγο πολύ. Τα υπόλοιπα δεν έχουν υπαχθεί σε δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά πάλι είναι υλικό προς επαλήθευση. Έχουμε κάνει πολλές επαληθεύσεις οικονομικές, πολλές φορές έως και υπερβολικά, γιατί θεωρητικά θα έπρεπε το 7% των ε, δικαιούχων υπό το ορίζον 2020 να είναι το ελεγχόμενο, ελεγχόμενος πληθυσμός, αλλά έχουμε περισσότερο. Για τα καταποκοπήν ποσά. Είναι ξεκάθαρη κατάσταση από το ορίζον 2020, έχουμε ξεκινήσει από την αρχή, δεν υπάρχει ετεροχρονισμένος υπολογισμός. Πιστεύω ότι θα είναι σαφής η κατάσταση αν και δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα ακριβώς την ερώτησή σας, γιατί δεν βλέπω τι ακριβώς μπορεί να εννοείται ως ε, αναδρομικό υπολογισμό των καταποκοπήν ποσών, αν κατάλαβα καλά ότι αυτό ρωτούσατε. Η ερώτηση ήταν ποιο είναι το ποσοστό συνολικά των ποσών που έχουν καταποκοπήν καταβληθεί από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και άρα τι είδου επαληθεύσεις έχουμε στα καταποκοπήν ποσά, μέσα στην αναλογία μόνο των καταποκοπήν ποσών. Και το ρωτώ βεβαίω διότι από τον τύπο ακούμε ότι υπήρξαν κάποιες επαληθεύσεις δημοσιονομικές. Και αν ευσταθούν τα άρθρα αυτά, δημιουργηθεί ένα κλίμα δυσφορίας από πλευρά των δικαιούχων για τις απολυθέσεις αυτές. Μπορείτε να μας ε, απαντήσετε. Σε ό,τι αφορά τα καταποκοπή ποσά, γίνονται πολλοί υπολογισμοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό του καταποκοπή ποσού. Υπάρχουν ε, διαφορετικά ποσά για διαφορετικούς δικαιούχους. Δεν ξέρω πόσο είναι το εύρος. Και επίσης ε, τα καταποκοπή ποσά δεν υφίστανται λογιστικό έλεγχο. Ε, απλώς χορηγούνται. Τώρα θέλετε ποσοστά και ποσά. Θα μπορούσα να σας απαντήσω γραπτός βεβαίως. Πόσα, πόσα καταβάλλονται, ξέρω εγώ, 20%, 60% ε, στο ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7 και μαζί με τις υπόλοιπες ε, πληροφορίες για τις ε, υποθέσεις στην Όλαφ και την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Άνια δεν έχω πάθει ακόμα. Θυμάμαι τι σας έχω ρωτήσει και που μας έχετε τάξει απάντηση. Καλό θα ήταν να μας τη δώσετε για αυτή την απάντηση και σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η συγκήτρια για να ολοκληρώσει τότε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κρίμα που δεν προλάβαμε να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και το τόσο σύντομη συζήτηση. Θα εμβαθύνουμε επ' ευκαιρία των τροπολογιών και της εξέτασής τους. Θα καταθέσουμε τροπολογίες για την ελαστικότητα ευελιξία μεταξύ των προϋπολογισμών, μεταξύ των προγραμμάτων. Θα ζητήσουμε απλούστευση και καλύτερη καθοδήγηση των δικαιούχων θα θέλαμε επίσης καλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων στα προγράμματα αυτά. Αυτό το αντικείμενο θα έχουν οι δικές μου τροπολογίες και φαντάζομαι ε, θα επιμικηθεί κάπως το σχέδιο έκθεσης ε, με τη συμπερίληψη και των ε, τροπολογιών γιατί για το προκαταρκτικό σχέδιο έπρεπε να τηρήσουμε τους περιορισμούς για την έκθεση. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μας δώσατε και κατά την εκπόνηση του σχεδίου και σίγουρα θα επανέλθουμε με υποβολή νέων ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό της ημέρης της δέταξης. Επειδή έχουμε ορίσει ώρα ψηφοφορής την Τετάρτη απογευματινή, τίστε τώρα το ερώτημα, μπορούμε να ψηφίσουμε. Θα φέρετε οι πολιτικές ομάδες στον κόσμο σας εδώ για να ψηφίσουμε την ε, έκθεση που είναι σημείο 5 και η γνωμοδότηση του συναδέλφου Αλή. Μπορούμε να ψηφίσουμε πριν τις 4 ή πρέπει να ψηφίσουμε ακριβώς τις 4. Άρα ψηφίζουμε την ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Η κυρία Πιτέρα είναι η συγκήτρια μας. Das gut, wenn man zumindest mal eine Abstimmungsliste hätte. Και να είχαμε και κανένα κατάλογο ψηφοφορίας θα βοηθούσε τα μάλα. Λοιπόν, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο εξή. Όταν ψηφίσαμε την απαλλαγή ξεχάσαμε κάτι να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ε, προς το δικαστήριο. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν ήταν στον κατάλογο ψηφοφορίας και θα ήθελα ε, να ε, την ψηφίσουμε τώρα. Ορίστε τι θέλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να περιμένουμε πέντε λεπτά γιατί δεν είναι πλήρης η ομάδα μας ακόμα. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά διακοπή και αμέσω μετά ακολουθούν ψηφοφορίε. Πρώτα η γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γιούρη για την απαλλαγή του δικαστηρίου και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Ich sehe, Βλέπω να πυκνώνουν οι γραμμές σας και ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την απαλλαγή ε, του δικαστηρίου. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, εν μπλοκ. Διαφωνεί κανείς. Όχι. Διαφωνεί. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν Γιούρι 4, Γιούρι 6, Γιούρι 7 και Γιούρι 9. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα το σύνολο. Ωραία. Το διεκπαιρεώσαμε και αυτό και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Πιτέρα. Δεν ξέρω, θέλει συγκίτρια το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι άλλαξα ε, σύσταση ε, σε ό,τι αφορά την τροπολογία 5 της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Άλλαξα γνώμη αφού ανέλησα την τροπολογία αυτή. Παρόλο που είχα βάλει αρχικά θετικό πρόσημο, προτείνω να βάλουμε ανετικό. Ευχαριστώ πολύ. Στη σελίδα 3 θα βρείτε την τροπολογία αυτή. Παράγραφος 8β νέα. Λίμπε 5, μάλιστα. Είναι τεράστια η προσψηφοφορία. Αρχίζουμε συμβαστική 1. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 32 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 33 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Σε διατμήματα τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία του αριθμού 37 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Η 42 υπέρ. Κατά. αποχέ. απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Χρειάζεται ηλεκτρονική επαληθεύση παρακαλώ για τις 40 ενέργειες τώρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. 51 υπέρ. Δεν καταπέφτει 50. Όχι, όχι. Όχι. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ καταπίπτει μάλλον. Ζητώ συγγνώμη. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 8 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να την ελέγξουμε, Ρέτζι 8, παρακαλώ.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 97 εφέ κατά αποχές εγκρίνεται 98 εφέ κατά αποχές απορρίψεται 99 εφέ κατά αποχές εγκρίνεται 100 εφέ κατά αποχές εγκρίνεται 101 καταπίπτει 102 επέ κατά αποχές απορρίψεται 103 επέ κατά μπορούμε να την ελέγξουμε την 103 παρακαλώ Πέρας. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. 110. Κάποιοι συνάδελφοι δεν σηκώνουν χέρια. Πέρας. Απερίφθη. 111 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Τι θέλετε να ελέγξουμε την 112. Ήταν υπέρ. Εγκρίθηκε, σαφές. Πέρασε. 113 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 116 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 117 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 Πρώτο τμήμα. Πόσα τμήματα έχει εδώ? Α, το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα τώρα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 164 καταπίπτει, 166 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 165 και 167 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 168 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέ. κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 καταπίπτει 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 καταπίπτει 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέγγι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 9. Check Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 επε κατά αποχές απορρίπτεται 20 επε κατά αποχές απορρίπτεται 22 επε κατά αποχές εγκρίνεται 23 επε κατά αποχές εγκρίνεται 24 επε κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 1 μέχρι και 11 έχει καλυφθεί, Λίμπε ε, έχει καλυφθεί όλες οι τροπολογίες ε, και όλη η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελευθεριών καλύπτεται και δεν ψηφίζεται, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια. Γιούλια Πιτέρα. Right. Thank Σας ευχαριστώ λοιπόν. Περνάμε στην έγκριση του σχεδίου έκθεσης ε, για την ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ για το 2015. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Άλλη. Μήπως θέλει το λόγο? Θα ήθελα Απλώς να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα. Παρά τα προβλήματα που είχαμε αρχικά, τελικά η επικοινωνία αποκαταστάθηκε και το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, είναι ικανοποιητικό. Αυτά, ευχαριστώ. 184 τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά yeah. I'm sorry. I would like to have a voting list as well from my own group. That's why then I can better see. Δώστε μου τον κατάλογο ψηφοφορίας ε, από την ομάδα μου για να διαπιστώνω ε, που κυμαίνεται η πλειοψηφία, γιατί έχασε τη δικιά μου. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές.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 αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 12 άρχεται ψηφοφορία. Πέρα στο ελέγχο εγκρίνεται. Τροπολογία 13 καταπίπτει. Η 14 το ίδιο και πάμε στη 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 και 18 μαζί και 17 λιπρόδες, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ,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 Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 27. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το εξακριβώσουμε με τον έλεγχο. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Ναι, ναι, ναι, με φανή διαφορά. Τροπολογία 28. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά αποχές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 33 καταπίπτει, 34 το ίδιο, 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 39 καταπίπτει, 40, 40-42 καταπίπτουν, 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Η 57 κατά 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές, απο... ή μάλλον εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται, λέει η 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 καταπίπτει. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 86, αν και μάλλον εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 και 108 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 καταπίπτει. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 117 που μάλλον εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές ...128 μάλλον πρώτα, υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 128, άρχεται η ψηφοφορία. And it is rejected απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 131. Checks over. Απερίφθη. Εκατόν τριάντα τρία. Εκατόν τριάντα δύο. Εκατόν τριάντα δύο υπέρ. Κατά. Αποχές να το επαληθεύσουμε. Πέρασε εγκρίνεται 134 υπέρ 133 μάλλον πρώτα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 139 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 140 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 141 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε το 145. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. 145. Απεριφθεί όντως. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά 147 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. 147 απερίφθη 147 και πάλι 148 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 151 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 153 κατά πίπτη 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. 154. Και πέρασε. Απερίφθη. 155 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 155. Επαληθεύουμε. Πέρασε. Απερίφθη. 156 υπέρ κατά αποχές. 156. εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 159 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 160 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 162 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 166-167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 169 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 177 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 178 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 181 υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθη, 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Οι 4 της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής εγκρίνεται, να τις κάνουμε μέχρι τις 12, από την 6 μέχρι τις 12 της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. On block, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνονται το σύνολο Το σχεδίου ονομαστικά. Πέρας. 16 υπέρ, μία ψήφος κατά και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σπουδαίο νομοθέτημα. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και περνούμε στο σημείο 7, 8, συγγνώμη, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα ο εισηγητής ε, για το 7ο. Λοιπόν, έχουμε την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. κανόνες περί ενισχύσεων, πολιτικής συνοχής, με τον συνάδελφο Αλή εισηγητή, τον κύριο Χέριξ από το ελεγκτικό συνέδριο. Καλώς ήρθατε. Είστε στην ηλιόλουστη πλευρά της ζωής καθισμένος. Παρακαλώ λοιπόν για να, κάνουμε, να δούμε την παρουσίαση. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τις κύριες διαπιστώσεις και συστάσεις τη έκθεσή μας για τις κρατικές ενισχύσει τη πολιτική συνοχή, Ξεκινώντας όμως θα ήθελα να σας πω μια γενική, να μια γενική διαπίστωση ότι κατά βάση και γενικώ υπάρχει απαγόρευση από την ε, συνθήκη για τις κρατικέ επιδοτήσεις και βέβαια υπάρχουν και τομεακέ διευκρινήσει και γεωγραφικές. Για την περίοδο 2007-2013 το συνολικό ποσό των κρατικών ενιστοιχήσεων ήταν 504 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 139 δισεκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο για την Πολιτική Συνοχής. Ελέγξαμε λοιπόν το βαθμό μη τήρησης των προδιαγραφών των σχετικών με τις κριτικές ενισχύσεις. Μετά τις διαπιστώσεις των παραβιάσεων είτε από το ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή ή τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια κάναμε την ανάλυση των σφαλμάτων και των διορθωτικών μέτρων που έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διορθωτικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 και τις δράσεις που έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινούμε λοιπόν με τις κύριες ε, διαπιστώσεις μας. Έχουμε περίπου ποσοστό σφάλματος 13,5% με αναλογία για την περίοδο 2010-2014 για την πολιτική συνοχής σε επίπεδο 5,7% σημαντικός μονοτομέας, αλλά υπάρχει πάλι υπάρχει τάξη μεγέθους. Έχουμε ως ε, σφάλματα το ύψος της ε, κρατικής ενίσχυσης ε, και άλλα ζητήματα. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Απασχόλησης και άλλες έχουν εντοπίσει σφάλματα, αλλά δεν τα έχουν ε, αναλύσει επαρκώς και άρα είναι ελλειπής η ανάλυση και η συμπλήρωση των βάσεων δεδομένων. Δεν μας επιτρέπουν δηλαδή να αναλύσουμε πιο σωστά την κατάσταση και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει εισαγάγει πολύ πιο στοχευμένα μέτρα και προληπτικά μέτρα για τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν συνέβη λοιπόν η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό από την άλλη έχει προβεί σε μια οριζόντια ανάλυση επί τη βάση των ε, εποπτευωμένων ε, κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2006-2014, ανάλυση η οποία δίνει ως αποτέλεσμα ένα 30% των ενισχύσεων ως προβληματικές. Αυτές καταχωρούνται λοιπόν ως προβληματικές που σημαίνει ότι ε, παραβιάζουν κάποιες διατάξεις σχετικές με τον ανταγωνισμό πιο συγκεκριμένα κράτη-μέλη, πέντε συγκεκριμένα κράτη-μέλη παρουσιάζουν ποσοστό ε, προβληματικών ε, περιπτώσεων ή ε, περιπτώσεων στις οποίες έχουν εντοπιστεί σφάλματα 50%. Στη συνέχεια βλέπετε μια πιο ακριβή ανάλυση της διάγνωσης φάλματος στην διαφάνεια αυτή το ελεγκτικό συνέδριο έχει ένα, 90, ε, ένα 19 περίπου της 100 εντοπίσει ε, ως ε, περιπτώσεις που παρουσιάζουν σφάλματα. Αντίστοιχο ποσοστό με αυτό της Γενικής Δεύτερης Περιφερειακής Πολιτικής από τις δικές της επαληθεύσεις και τους ελέγχους. Ενώ η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό έχει εντοπίσει παρατυπίες μέχρι ύψους 36%. Ε, βεβαίως αυτό θα εξηγηθεί και από διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχουμε, είτε δειγματοληπτικού ε, δειγματοληπτικούς ελέγχους, είτε ε, προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο που έχει η τον ανταγωνισμό. Σημαντικό πάντως βήμα έχει πραγματοποιηθεί προς, την, προς τη διαπίστωση αυτή και τον συντονισμό. Τα κράτη-μέλη έχουν ποσοστό χαμηλότερο από 4% σφάλματος εντοπίσει. Δηλαδή, πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με διαφορετική και πιο συστηματική διερεύνηση έχουμε ποσοστό έως και πενταπλάσιο από αυτό των κρατών μελών εντοπίσει. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη στι ε, επαληθεύσει και του ελέγχου του δεν, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στι κρατικέ ενισχύσει. Εντοπίζουμε ω πρόβλημα τον ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ Επιτροπή ε, δεν υπάρχει δηλαδή ανταλλαγή ευρημάτων και αναλύσεων μέσα μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Η μία έχει πολύ περιορισμένο η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μιας άλλης γενικής διεύθυνσης και ούτω καθεξής. Επίσης, προγράμματα με κόστος των 50 εκατομμυρίων ευρώ δεν υπάγονταν σε συστηματική απαλήθευση από τις Γενικές Διευθύνσεις ε, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανταγωνισμού ε, πριν από την υπόθεση Leipzig Χάλε του 2012. Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να εγκρίνονται μεγάλη κλίμακας έργα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση των διατάξεων περί ε, κρατικών ενισχύσεων και άρα να παρεμβάσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από το 2007 το τέλος του 2012 σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκραίνει 440 μεγάλης κλίμακας έργα και πολύ λίγα από αυτά έχουν κοινοποιηθεί. Επίσης επιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ λίγα διορθωτικά μέτρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάλι σε αναλογία των σφαλμάτων που έχουν εντοπίσει οι δύο γενικές διευθύνσεις. Από την Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση έχουμε 18 δημοσιονομικές διορθώσεις για τα κράτη-μέλη στην περίοδο 2010-2014, αυτήν την πενταετία, με 59 περίπου εκατομμύρια ευρώ χρηματοοικονομικό όγκο, αντίστοιχο με αυτόν των κρατικών 95 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό έχει σε μία μόνο περίπτωση κάνει διορθωτική, ε, διόρθωση χρηματοοικονομική, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό δηλαδή διόρθωσης για την ε, προγραμματική περίοδο 2014-2020. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Εδώ έχουμε το γενικό κανονισμό Τζίμπερ ενισχύει πλέον που ενισχύει σημαντικά, διευρύνει σημαντικά το πεδίο και βλέπουμε ότι 70% των κρατικών ισχύσεων καλύπτονται από τις λεγόμενες εξαιρέσεις. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη σε επίπεδο κρατών μελών πλέον, τα οποία καλούνται να εντοπίζουν το πρόβλημα. Άρα ε, ενισχύεται το δυναμικό κινδύνου να προκύψουν προβλήματα τα οποία τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταγράψει. Κράτη-μέλη τα οποία έχουν δηλαδή διαπράξει σφάλμα σε σχέση με, τη, το γενικό κανονισμό καλούνται να βελτιώσουν τα ποσοστά διόρθωσης. Έχουν εντωμεταξύ για την περίοδο 2014-2020 βελτιωθεί οι συνθήκες για τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις και για την προσαρμογή τους για το καθεστώς των ενισχύσεων που πηγαίνει πάνω από τα 500.000 ευρώ και παίρνω πολύ γρήγορα στην περιγραφή άλλων νέων στοιχείων του καρονισμού ή εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για, την, για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα κράτη-μέλη προβαίνουν σε μια αυτοαξιολόγηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πέντε κράτη-μέλη φάνηκε ότι οι συνθήκες αυτές ε, που προβλεπόταν για την έγκριση, προβλέπονταν για την έγκριση των εταιρικών σχέσεων δεν πληρούνται. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε πρωτοβουλίες που ονομάζονται σχέδια δράσης σε σχέση με τα κράτη αυτά, εκ των οποίων εντωμεταξύ το ένα έχει κάνει τη σχετική διόρθωση. Έχει ξεκινήσει λοιπόν πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα κράτη-μέλη για να βελτιώσει και το διοικητικό δυναμικό των ε, κρατών μελών με την κατάρτιση, καλύτερε βάσει δεδομένων καθεξής. Θετικά μέτρα τα οποία θέλαμε να ε, επισημάνουμε και για να φτάσω στι συστάσει μας πολύ συνοπτικά. Έχουμε 12 επιμέρους συστάσεις, διατυπώσει. Με αποδοχή από πλευράς της Επιτροπής του μεγαλύτερου τμήματος, εκτός από τρεις η βελτίωση της επιτήρησης του follow-up από πλευράς Ευρωπαϊκής είναι η κυριότερη σύσταση. Θα πρέπει να αξιοποιεί δηλαδή και τη βάση δεδομένων και όλα τα στοιχεία που είστε θέσει της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εντοπίσει αλλά και να αναλύσει καλύτερα το είδος, ε, την πυκνότητα, τη συχνότητα ε, και το ειδικό βάρος των σφαλμάτων και παράλληλα να ε, παρακολουθεί τα κράτη-μέλη ώστε να τους συνιστά τις διορθώσεις και διορθωτικά μέτρα εάν δεν είναι ε, ικανοποιητικά τα διορθωτικά μέτρα σε σχέση με τις ε, προδιαγραφές για τις κρατικές ενισχύσεις. Μεγάλα έργα λοιπόν μπορεί να εγκρίνονται με βάση και τις διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις εφόσον έχουν υλοποιηθεί ε, μεγάλου όγκου και ικανοποιητική ποιότητα επαληθεύσει και από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει συγκεκριμένους δείκτες και με παραδείγματα ακόμη να καθοδηγεί τα κράτη-μέλη ώστε ε, να αντιμετωπίζονται, να προλαμβάνουν αυτά τα σφάλματα και μάλιστα θα μπορούσε να δώσει και συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχει ένα είδος σφάλματος το οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί σε μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με βάση την αρχή Ντέγκεντορφ για να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να καταγράφουν ε, τις ε, ε, ενισχύσεις έστω με, με τον καρόνα Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με στη θέση σας για ερωτήσεις. Äh, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εντυπωσιακή ειδική έκθεση. Ε, για κάποια θέματα που μέχρι τώρα δεν τα είχαμε, δεν τους είχαμε δώσει τη σημασία που επιβάλλεται. Ο συγητής, ο κύριος Αλή, παρακαλώ. Αγαπητέ ε, κύριε Χέρεξ, Κυρίες και κύριοι, πάνω από ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για τη διαρθωτική πολιτική, οικονομική, πολιτική, οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή. Επαναβιομηχάνηση, ε, και ενίσχυση της γεωργίας εκεί που παρακμάζει. Άρα θα πρέπει οι περιφέρειες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να αναπτυχθεί η οικονομία τους και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις απαγορεύονται για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, σε ειδικού τομεί, σε συγκεκριμένε γεωγραφικέ περιφέρειες και μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό μπορεί αυτέ να επιτρέπονται. Στόχος του ελέγχου ήταν να εντοπιστούν οι περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες και σε ποιες περιπτώσεις έχει ε, λάβει γνώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μη συμμόρφωση έτσι ώστε ε, να σχεδιαστούν δράσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο έκανε μια εξαιρετική ε, εκτίμηση και έλεγχο στην προγραμματική περίεργο 2007-2013 με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο 2010-2014. Η ειδική έκθεση επίσης αναλύει κατά πόσο η δράση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει και σε σχέση με ε, τη δυνατότητα των κρατών μελών να βελτιώνουν τις επιδόσεις και να ελέγχουν ε, τις παραβιάσεις και παραβάσεις για να έχουμε μία αξιόπιστη εικόνα του τι συμβαίνει στην πολιτική συνοχή, να χαραχθούν κατευθυντήριε γραμμέ ε, σωστέ για το μέλλον. Είμαι επίση ικανοποιημένο από την απάντηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ειδική έκθεση, ιδιαίτερα από την προθυμία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, δεχθεί τι περισσότερε ε, συστάσει. Κάποιε από αυτέ μπορεί να συζητηθούν περαιτέρω, πάντω γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνη. Ε, έτσι ώστε να αποτρέπονται και να προλαμβάνονται παραβιάσεις ε, των κανόνων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί συζήτηση. Και αν δεν συζητούσατε και κοιτούσατε όλοι τα mail σας τώρα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια σημαντική έκθεση. Οι ε, πάντες κοιτάνε τα mail τους. Καλώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Γενική Διεύθυνση Ρέτζι και ε, ανταγωνισμού και από την Όλαφ. Ποιος θα αρχίσει. Many uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας είμαστε ευγνώμονας και ιδίω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτή την ε, ευρυθή ανάλυση. Έχουμε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για να εντοπίσουμε τα θέματα και να τα διαλευκάνουμε ως προς τις κρατικές ε, ενισχύσεις και όχι μόνο εν ώψη αυτής της ε, ειδικής έκθεσης, γιατί και με την δήλωση των ΤΑΣ από το 2013 και 2014 ήδη είχαμε επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα των κρατικών ενισχύσεων που ήταν από τις βασικές πηγές φάλματος στην Επιτροπή Συνοχής μεταξύ 17 και 20% του ποσοστού σφάλματος. Είμαστε ευγνώμονες προς το ελεκτικό συνέδριο για την ανάλυση που μας έκανε και επίσης αναγνώρισε το ελεκτικό συνέδριο ότι ε, μετά την πρώτη περίοδο ελέγχου το τόνισε ο κύριος Αλή, στην περίοδο δηλαδή κυρίως 13 με 14 διαπίστωσε ε, πρόοδο, βελτίωση. Είδαμε στην ε, της έκθεση του 2015 ότι τα θέματα κρατικής ενίσχυσης είναι 5,8% του ποσοστού σφάλματος και επίσης ε, το ελεκτικό συνέδριο στην ηθική έκθεση αλλά και στην ετήσια έκθεση για το 2015 διαπίστωσε βελτιώσεις στο έργο των ελεκτικών αρχών και στους ελέγχους που έκαναν σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. Είναι πρόσδεκτη αυτή η βελτίωση. Επίσης δεχτήκαμε εννέα συστάσεις, ε, τις ε, επεξεργαζόμαστε και μάλιστα το ελεκτικό συνέδριο αναφέρεται και ε, στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, στην οποία συμμετέχουν οι Γενικές Διευθύνσεις Ρέγγιο, Απασχόλησης και ανταγωνισμού προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν θέματα κρατικών ενισχύσεων που είναι αρκετά περίπλοκα. Εμείς έχουμε συνεργαστεί με τις, ε, αρχές, ε, τις Εθνικές Αρχές Ελέγχου για να βελτιωθεί η διοικητική τους ικανότητα και από το 2011 και πάλι ε, στο 2015 είχαμε λεπτομεριακούς καταλόγους προκειμένου, καταλόγους στοιχείων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τον έλεγχο και μάλιστα ενθαρρύνουμε τις αρμόδιες κρατικές αρχές να συμπεριλάβουν αυτούς τους καταλόγους με τα στοιχεία που θα πρέπει να ελέγχουν, ώστε να έχουμε σε ομοιόμορφα πρότυπα και προδιαγραφές στον τομέα αυτό διενέργειας ελέγχου. Επίσης, αναθεωρήσαμε και τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούσαμε για την ε, ενημέρωση θέματα μη συμμόρφωσης με θέματα κρατικών ενισχύσεων και από το 2013 είχαμε βάση δεδομένων, αλλά δεν ανταποκρινόταν ε, στο στόχο μας, δηλαδή στην εκπόνηση τέτοιων αξιολογήσεων που μας ζητά το ελεκτικό συνέδριο. Και για το επόμενη περίοδο προγραμματισμού μέχρι το 2020 θα έχουμε πολύ βελτιωμένα συστήματα και μια κατάλληλη βάση δεδομένων για να ε, ενημερώνει για ατασταλίες σε θέματα αυτά και για την τυπολογία του σφάλματος προκειμένου να ε, κοινοποιείται στις αρμόδιες ε, γενικές διευθύνσεις και στην ΟΛΑΦ αλλά και στους ε, αρμόδιους φορείς ελέγχου που ενθαρρύνονται σε αιτήσει εκθέσεις ελέγχου να μας ενημερώνουν για τα είδη σφαλμάτων και για την τυπολογία τους. Και ευελπιστούμε ότι αυτά τα νέα στοιχεία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερες αξιολογήσεις και να συνεργαστούμε με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τα πιο συχνά ασφάλματα, προκειμένου να έχουμε πιο στοχευμένες δράσεις στο μέλλον, σε περίπτωση που επαναλαμβάνονται συγκεκριμένα είδη ασφαλμάτων και όπου η συχνότητά τους είναι αυξημένη. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για να ε, σχολιάσει συγκεκριμένα θέματα αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσής του. Πάντως, ε, σε ό,τι αφορά την έκκληση του εισηγητού να αναθεωρήσουμε ή να παρήψουμε τη σύσταση, της 4 4β που αφορά κυρίως τα μεγαλεπίβολα, τα μεγάλες κλίμακα σχέδιων υποδομής που υιοθετήθηκαν πριν το 2012. So, όπως αναφέρεται και στην ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδριού, το 10 είχε συγκεκριμένη νομολογία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων σε σχέδια υποδομής, στα σχέδια υποδομών. Με την ομολογία αυτή διευκρινίστηκε κάπως ένας τομέας που ήταν κάποιος, κάπως ασαφής και ενημερώσαμε για τα κράτη-μέλη. Τέτοιου είδου ε, προγράμματα υποδομών δεν υπάγονται στου κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει. Με τη νέα νομολογία του ΔΕΚ του 2011, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη-μέλη ότι εξαιτία ε, τη νέα νομολογία θα έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση για αυτά τα μεγάλη κλίμακα σχέδια υποδομών και να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιθανά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο. Επίσης, ε, ε, εγκρίναμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές που στείλαμε σε όλε τις αρμόδιες ελεκτικέ αρχές και σε αυτές τις ε, κατευθυντήρες γραμμές από το 2012 διευκρινίζουμε ότι το αίτημα αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων για μείζωνα προγράμματα υποδομών μετά το 2012 ισχύει, γιατί δεν μπορούσαμε αναδρομικά να επιβάλλουμε κάποιες νομοθετικές διευκρινήσεις στα κράτη-μέλη ή να πλήξουμε τους δικαιούχους. Τους δικαιούχους. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο ε, που θα εξασφαλίζει σαφήνεια και για τα κράτη-μέλη και για τους δικαιούχους και, και αυτό με τις κατευθυντήριες γραμμές μας ε, δίνουμε σαφείς οδηγίες στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν μείζωνα και ε, μικρότερης εμβέλειας ε, σχέδια υποδομών και πριν αλλά και κυρίως μετά την υποβολή των κατευθυντηρίων γραμμών μας. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο τώρα να επανέλθουμε στο τέλος περίοδου προγραμματισμού, τώρα που θα, θα ολοκληρώσουμε αυτή την περίοδο προγραμματισμού την επόμενη εβδομάδα και τώρα ξαφνικά να πούμε στους δικαιούχους ότι αναθεωρούμε κάποιες υποθέσεις. Και μάλιστα, μια και ο κίνδυνο είναι περιορισμένο, όπω σα εξηγήσει και ο συνάδελφο, δεν κρίναμε ότι κάτι τέτοιο ήταν σκόπιμο ή απαραίτητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, βελτιώσαμε την διαδικασία έγκριση ε, σχεδίων μεγάλη κλίμακα ε, ώστε να διευκρινιστεί οποιοδήποτε θέμα κρατική ενίσχυση μεταξύ του κράτου μέλου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα πριν την υιοθέτηση ε, οποιασδήποτε απόφαση ε, για έγκριση μείζωνο σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε έχουμε ε, αυστηρότερη διαδικασία για την περίοδο 2014-2020 και θα πρέπει να διευκρινιστούν οποιαδήποτε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων πριν τη λήψη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν έχει νόημα να εγκρίνουμε ένα μείζον σχέδιο υποδομής και κατόπιν να ενημερώνουμε το κράτος μέλος ότι δεν ήταν τελικά επιλέξιμο. Επίσης είχαμε στενή συνεργασία με τις ελεκτικές αρχές των κρατών μελών για να ενισχύσουμε, να την ικανότητά τους. Και δεν μιλώ για μόνο για καθοδήγηση, ε, κατάρτιση ε, επιτόπου, εκπαίδευση και τον κατάλογο αυτό με τα στοιχεία που θα πρέπει να τσεκάρουν τα κράτη-μέλη, αλλά ενημέρωση και για την ομολογία και μάλιστα στην ετήσια έκθεση ελέγχου του 2015 το ελεκτικό συνέδριο ε, διαπιστώνει βελτιώσεις στους ελέγχους που διεργούν οι εθνικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με προηγούμενες χρόνιες. Και μάλιστα οι περισσότεροι έλεγχοι που γίνονται χάρη στους καταλόγους αυτούς με τα στοιχεία που θα πρέπει να ζεκάρουν έχουν εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμόρφωση με θέματα κρατικών ενισχύσεων οπότε διαπιστώνεται σχετική βελτίωση από το ελεκτικό συνέδριο. Πάντω συνεχίζουμε τη συνεργασία με τι ελεκτικέ αρχέ και τι αρχέ ε, προγραμ... Ε, διαχείρισης προγραμμάτων και με το τρέχον σχέδιο δράση. Έχουμε βελτιώσει κατά πολύ τη συνεργασία και το συντονισμό και με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τα θέματα αυτά και ε, συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη προκειμένου να αποκαταστήσουμε πλήρη διαφάνεια, ε, σαφήνεια μάλλον, σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόμπερ. Δεν αντελήφθη γιατί δεν έχει προβεί σε διορθωτικά μέτρα μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήταν χρήσιμε οι στάσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Ποιο θα λάβει το λόγο μετά από εσά. Εξηγήστε πρώτα εσεί Σύσταση παριθμών 1. Αυτή αναφέρεται, αφορά κυρίως την ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Αλλά κυρία Πρόεδρε, το ελευθερικό συνέδριο αναφέρεται στην ε, διάγνωση και τη διόρθωση από πλευράς της Γενικής μας Διεύθυνσης σε όλες τις περιπτώσεις ε, παραβίασης των αρχών περικρατικών ενισχύσεων και διαπιστώνει ότι έχουμε επίπεδο διορθώσεων αντίστοιχο με αυτό του ελευθερικού συνεδρίου ως Γενική Διεύθυνση και νομίζω ότι αναφέρθηκαν από το Ελεκτικό Συνέδριο 7 κρατημέλη στα οποία έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορθώσει διορθώσεις ε, οικονομικές λόγω της ε, διαπίστωσης του σφάλματο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την παρακολούθηση λειτουργίας των ε, προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. για τις τρεις συστάσεις που απέριψε η Επιτροπή, ήθελα να αναφερθώ. Αλλά μια και μιλήσατε για τη διόρθωση σφαλμάτων από την επιτήρη, που διαπιστώνονται στην επιτήρηση. επιτρέψτε μου δύο λόγια σε αυτό. Λοιπόν, όντω έχουμε τέτοιου είδου ζητήματα κάθε χρόνο, με ένα επίπεδο περί το 30% διόρθωση ε, σφάλμα, μάλλον διάγνωση σφάλματος. Το σφάλμα όμως δεν σημαίνει ότι είναι ασύμβατες ε, οι κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ παρατυπίας της ενίσχυσης, δηλαδή ότι δεν είχαν τηρηθεί οι όροι ε, συμμόρφωσης και ασυμβίβαστου που είναι ε, παραβίαση σε σχέση με την ουσία. Επίσης πολύ συχνά έχουμε προβλήματα τήρησης των διαδικασιών από τα κράτη-μέλη. Και άρα δεν είναι πάντοτε ουσιαστικά τα προβλήματα παραβίασης της, ε, ε, του ασυμβίβαστου, ε, της ουσίας. Τα διαδικαστικά ζητήματα μπορούν να αφορούν νομική βάση που προβλέπει μια σειρά από προϋποθέσεις και που ίσως εκ πρώτης όψης να φαίνεται πως αντιρρήθηκε, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεται πως ε, υπάρχουν, ε, συντρέχουν όλοι οι όροι της νομικής βάσης. Και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να κάνει τις διορθώσεις και τις ε, διαδικαστικές. Εάν όμως δεν συμβεί αυτό, προχωρούμε σε ανάκτηση. Αυτό θα σας εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ ποσοστού σφάλματος και ανάκτησης, ανακτώμενων ποσών. Επίσης πολλές φορές με, την, ε, με τις διαπιστώσεις σφάλματος ε, γίνεται ε, εθελοντική ανάκτηση και έτσι δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καν να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκτησης και να πιέσει τα κράτη-μέλη για την επιστροφή των ποσών. Για τις τρεις συστάσεις Πρώτον, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει έργα που έχουν να κάνουν με ενισχύσεις πριν από, τις, από τη δίκη Λάτσι Χάλε. Κοιτάξτε, στην υπόθεση αυτή υπήρχαν ζητήματα που δεν είχαν εκριθεί μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ε, οι προσφερόμενες υποδεμές, επενδύσεις σε υποδομές θα μπορούσαν να κρυθούν ως κρατικές ενισχύσεις. Ε, αυτό έμενε αστροφές και το διευκρινίζει με την απόφαση του το δικαστήριου στην απόφαση Λάψη Χιάλα. Έτσι λοιπόν αυτούς τους καρόνες όπως διευκρινίστηκαν μπορούμε να τους ελέγξουμε ε, στο μέλλον. Αλλά δεν μπορούμε αναδρομικά να επικαλεστούμε παραβίαση κανόνων. Επίσης, στην έννοια της ενίσχυσης με την απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πέρσι, ε, δηλώνεται ότι η απόφαση Λάτσι Χάλε δεν λέει ότι κάθε είδους επενδύσει σε υποδομές μπορεί να είναι κρατικές ενισχύσεις. Ε, κρίσιμες υποδομές, σιδηροδρομικές γραμμές, οδικές αρτηρίες, ε, παροχή ύδατος κτλ. δεν υπάγονται στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης. Και έτσι σε τέτοιου τομεί μπορεί να αναπτύσσονται έργα τα οποία δεν καλύπτονται από τους όρους της κρατικής ενίσχυσης. Από την άλλη βέβαια ε, λιμενικές, αερολιμενικές εγκαταστάσεις και άλλες που μπορεί να εκτίθενται και σε περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ δικτύων, ε, ε, τότε ναι μπορεί να θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις. Άρα είναι περιορισμένο το πεδίο της αποφάσης Leipzig-Harlem και για, το, για την περίοδο πριν από την απόφαση, δεδομένου ότι δεν ήταν σαφής η κατάσταση και οι κανόνες, θεωρούμε ότι θα ήταν δι, διοικητικά κακή διαχειριστική πολιτική να ε, κοιτάξουμε αναδρομικά τις αποφάσεις, τις παλαιότερες. Επίσης, ε, κοιτούμε τα όρια τα οικονομικά των ποσών τα συνολικά να αξιολογούνται σε τριετία, δηλαδή σε μια περίοδο τριών ετών ποιο είναι το ποσό το οποίο έχει ε, λάβει μια επιχείρηση αν μπορεί να κρυθεί κρατική ενίσχυση. Αλλά όπω, είπαμε ε, δεν ε, διαπιστώνονται όλα τα προβλήματα μόνο από του δικού μα ελέγχου, Μπορεί και με αυτό δηλώσεις ή δηλώσει δηλώσεις τα κρατημέλη να προβαίνουν σχετικέ διορθώσει Και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε λύσεις ε, που ανέχονται και διαφορετικές μεθόδους από τα κράτη-μέλη. Επίσης, κεντρικό μικρό για τις εντολές ανάκτησης. Η απόφαση Technicourt πριν από μερικά χρόνια είχε δώσει την... Ε, η απόφαση Technicourt είχε δώσει το τεχνικό στοιχείο του τι μπορεί να ε, χαρακτηρίσει κρατική ενίσχυση. Είπαμε ότι η απόφαση αυτή, η απόφαση δεν αφορά μόνο αρχικό επίπεδο. Η νέα ενίσχυση πρέπει να ε, διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο και με βάση τον κανονισμό θα υιοθετηθούν νέες διατάξεις. Ένα ενοποιημένο λοιπόν μητρό με όλες τις νέες επιχειρήσεις δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τις ε, ε, στο σημείο αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν για την τήρηση των όρων του Ευχαριστώ. Η πρόσωπο της Όλαφ, ε, ζητώ συγγνώμη για το όνομα σας, Μαρία Σιγιουτούμα. Θα είμαι σύντομη σε ό,τι αφορά ε, τη σύσταση για το σύστημα διαχείρισης τη τη συμμόρφωσης 2β ε, και ΣΥ. Ήδη έχουμε υλοποιήσει εμεί τη σύσταση αυτή. Όπως είπε και ο κύριος Σίμπερ, έχουμε μια κοινή ε, μορφή διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων και των ελέγχων αυτό στο σύστημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είδατε, όταν δουλεύουν όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Κύριε Χέριξ, ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε, όσο και αντιφατικές ορισμένε απόψει, αντικρουόμενες μάλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τι θα λέγατε, πώ θα τα σχολιάσετε όλα αυτά. Έχετε το λόγο. Α, ζητώ συγγνώμη, κύριε Χέριξ. Κύριε Χέριξ, Äh, Kommission. ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Για τη σύσταση 4β, ε, ίσως κάποια τεχνικά να πω για κάποιες περιπτώσεις που εγκρίθηκαν πριν από το 2012, κατά πόσο αυτές θα πρέπει να επανελεγχθούν. Σας ανέφερα κάποια αριθμητικά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 440 έργα μέχρι το 2012, από το 2007. Και αν δούμε τις περιπτώσεις που κοινοποιήθηκαν, εγώ στατιστικολόγος δεν είμαι, από την ειδική έκθεση για την ε, αντίστοιχη περίοδο, ε, ήταν πολύ λίγα τα έργα που κοινοποιήθηκαν και εδώ υπάρχει μια μαύρη τρύπα, μια μάζα που δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και μπορούν να υπάρχουν σημαντικές παραβιάσεις ή ε, ανακτήματα για ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς απλώς να το επισημάνουμε θέλαμε. Μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει και η ζωή συνεχίζεται ή ασχολούμαστε με τη διερεύνηση και τη διελεύκανση αυτών των ε, υποθέσεων. Πρέπει να πω ότι κατανοώ το ε, τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω ασχοληθεί επανειλημμένα με τις κρατικές ενισχύσεις. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις του δικαστηρίου ε, στο... στη σελίδα 38 ε, το Δεκέμβριο του 2020 για το αερολιμένα Aéroport την αντίστοιχη εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ με δική της πρωτοβουλία και αυτό το λέμε στη σελίδα 62 έχει εγκρίνει ε, κρατικές ε, ενισχύσεις, τις έχει κατατάξει ως τέτοιες. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι συνιστά αυτοκρατική ενίσχυση, μπορεί να συνιστά και να εγκρίνεται. Άρα ε, νομίζω θα ήταν σκόπιμο και δικαιολογημένο να διευκρινιστούν όλα αυτά πριν την τελική για τη συμβατότητα και τα όσα είπε πρόσωπο Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι γεγονό. Δεν σημαίνει κάθε σφάλμα ότι ε, χρειάζεται επιστροφή των, ε, αποκτηθέντων προς... Ε, ποσών. Και στη σελίδα 34 αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις οι οποίε είναι προβληματικές και στην τελευταία στήλη κατά πόσο αυτές συνάδουν με την εσωτερική αγορά και στη σελίδα 9 με 14 έχουμε 16 σφάλματα, αλλά και άλλα σφάλματα που είναι ασυμβίβαστα ε, με την εσωτερική αγορά και ασύμβατα. Και τα λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχει προβεί σε μία διόρθωση μόνο, Γενική Διεύθυνση ε, Ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις τρεις συστάσεις τις οποίες αναφερθήκατε, Πρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ανέφερα ήδη την περιπτωση Λάιπτσιχ Χάλε. Και ε, υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις προς άλλη κατεύθυνση για το de minimis. Μιλήσατε για ασφάλεια δικαίου. Θα μπορούσα να το επικαλεστώ και εγώ για τη συγκεκριμένη ε, σύσταση. Να υπάρχει ένα μητρό που μπορεί κανείς να ελέγχει τι έγινε. Νομίζω στην Πορτογαλία υπάρχει μια αντίστοιχη υπόθεση και αυτό δίνει και προσδίδει ασφάλεια δικαίου. Ξέρετε ότι θα πρέπει να συναπολογίζονται ενισχύσεις τριών ετών για να δούμε αν έχει ε, ξεπεραστεί το όριο των 200.000 ευρώ. Και αυτό δίνει ασφάλεια δικαίου και δίνει και κάποια βεβαιότητα σε σχέση με το κόστος και την ωφέλεια. Και κάτι πρέπει να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθούν αυτή την οδό ή όχι. Και ε, ε, τη σχέση έχει η αρχή Ντέγκεντορφ, λέει ότι δεν μπορώ να δώσω κρατική ενίσχυση εφόσον εκκρεμεί επιστροφή χρημάτων από μια εταιρεία που πρέπει εγώ να τα ανακτήσω. Ε, αυτό μπορεί να λύνεται σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά εδώ ε, έχουμε ε, διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, σε πολλές χώρες, με ε, πολλές έτσι, νοοτροπίες και κουλτούρες διαφορετικές. Και για να έχουμε και εδώ μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου δεν θα πρέπει να εγκρίνονται, πόσο μάλλον να χορηγούνται ε, κρατικές ανισχύσεις σε εταιρείε από τις οποίες ζητούμε να επιστρέψουν ε, προς ανάκτηση ποσά. Ευχαριστώ, συνάδελφος Σάλα Φράγκα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή, το ελεκτικό συνέδριο, αλλά και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπαν που καταδεικνύουν μία από τις βασικές αρχές ε, των συνθήκων μας. Ε, η συνθήκη της Ρώμης κατοχυρώνει την ε, αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως θεμέλιο της εσωτερική αγοράς. Η ιδρυτική συνθήκη για την εσωτερική αγορά και που την εορτάσαμε την 60η επέτειο της εβδομάδας αυτής, της προηγούμενης μάλλον εβδομάδας, θα πρέπει να προβλέπει εύρυθμη λειτουργία και των, και των εθνικών οικονομιών. Δύο τρίτα της, των πολιτικών αφιερώνται στην πολιτική συνοχή. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μα δίνει το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί μα λένε τα στοιχεία αυτά ότι έχουμε 500 δισεκατομμύρια 500 δισεκατομμύρια περίπου κρατικέ ενισχύσει για αυτή την περίοδο. Είναι αστρονομικό το ποσό και 137 δισεκατομμύρια κρατικών ενισχύσεων που συνδέονται με την πολιτική συνοχή. Αυτά αποτελούν κατάφορη απόδειξη, άσχετα με την σκοπιμότητα τη έκθεσης ε, και την διεξαγωγή της συζήτησης, ότι 367 δισεκατομμύρια κρατικών ενισχύσεων αφορούν άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της πολιτικής συνοχής. Διαρωτώ με λοιπόν, γιατί ε, μόλις τώρα ανέλαβα τα καθήκοντα σε αυτήν την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Ε, είναι τεράστιο αυτό το ποσό, δεν είναι σκόπιμο να συζητήσουμε και για τις κρατικές ενισχύσεις ε, από άλλες ε, ευρωπαϊκές πολιτικές πριν της, πλην της πολιτικής συνοχής. Τώρα, συγκεκριμένη έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία και να ρωτήσω τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σφαλμάτων που έγιναν και του ποσού των ενισχύσεων που ανακτήθηκε. ανακτήθηκε. Από εκεί θα φανεί η αποτελεσματικότητα ή αναποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του συστήματο των κρατικών ενισχύσεων. Γιατί όπω είπα στην αρχή, δεν είναι εξορισμού παράνομε οι κρατικέ ενισχύσει. Είναι συμβατέ ή ασύμβατε με του στόχου τη συνθήκη. Θα ήθελα λοιπόν να με ενημερώσουν είτε εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου Ποια είναι η διαφορά σε απόλυτους όρους μεταξύ των σφαλμάτων που γίνονται στη, στις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει της πολιτικής συνοχής και τα επίπεδα ανάκτησης των αχρεωστήτων καταβληθέντων. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχθεί τις συστάσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου και ο εισηγητής το ίδιο. Οπότε Θέλουμε μια πιο ενημερωμένη βάση δεδομένων, κάτι που θα γίνει από ό,τι φαίνεται, και με καλύτερο συντονισμό όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά και μεταξύ των επιμέρους διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Γενικών Διευθύνσεων. Χρειάζεται ένα τέτοιο συντονισμό και εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη. Και τέλο, διάβασα με μεγάλη προσοχή το έγγραφο ε, εργασία του Ελεκτικού Συνεδρίου και με ανησυχία διαπιστώνω ότι πέντε χώρε μέλη δεν πληρούν τα κριτήρια για τα επίπεδα της ε, εκ των προτέρων ε, ε, υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχεδίων τους για τις κρατικές ενισχύσεις που θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια ως συμβατά ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να, γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη για να δούμε ποια είναι τα κριτήρια που δεν πληρούν το κριτήριο της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, γιατί είμαστε μια κοινότητα δικαίου και θα πρέπει να πληρούμε όλοι τις υποχρεώσεις μας στις ε, νομικές. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίες ερωτήσεις κύριε Ζέμπερ. Παρακαλώ θα μας απαντήσετε εσείς και οι συναδελφοί σας. Yes, Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Το ελεκτικό συνέδριο αναφέρθηκε στους υπολογισμούς που έκανε σε πέντε υποθέσεις, πέντε, για πέντε κρατημάλη σε σχέση με τις 18 υποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και αναφέρεται σε 36,8 εκατομμύρια διορθώσεις. Ε, από τα κράτη-μέλη, μόνο για τις υποθέσεις όμως που μπορούσε να συνδεθεί το θέμα της δημοσιονομικής διόρθωσης με την κρατική ενίσχυση. Και το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι μερικές διορθώσεις ε, δεν αφορούσαν τις κρατικές ενισχύσεις και γι' αυτό δεν μπορούσε να δώσει συγκεκριμένο στοιχείο για τις διορθώσεις που αφορούσαν μόνο κρατικές ενισχύσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημάνω εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε ξεχωριστά κάθε υπόθεση που φάνηκε στην έκθεση DAS ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου και επίσης παρακολουθήσαμε και τις ε, υποθέσεις που εντοπίσαμε εμείς και αυτές που μας ανέφεραν τα κράτη-μέλη. Και αυτό το αναφέρει στην ειδική έκθεση το Ελεκτικό Συνέδριο και εξηγεί ότι το επίπεδο ε, διορθώσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τις, είτε το, τη διάγνωση που έκανε το ελεκτικό συνέδριο της αναφοράς των κρατών μελών. Και όταν λέει το ελεκτικό συνέδριο στην ΤΑΣ ότι ένα σχέδιο ε, παρουσιάζει σοβαρές παρατυπίες ό,τι αφορά την ε, κρατική ενίσχυση και το ποσοτικοπίος 100% ε, σφάλμα ε, θα πρέπει εμείς να αξιολογήσουμε αν υπάρχει ε, ανάγκη κοινοποίησης ή όχι. Ακόμη και αν υπάρχει κοινοποίηση από το κράτος ε, μέρος στην περίπτωση αυτή, στη συνέχεια η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μπορεί να κρίνει ότι παρόλα αυτά η κρατική ενίσχυση είναι συμβατή με τη συνθήκη και την εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχει δηλαδή άμεσο σχετισμός μεταξύ του σφάλματος και συγκεκριμένη ποσότητα ε, και συγκεκριμένου ποσού, μάλλον που θα πρέπει να ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, υπάρχουν ε, πολλά είδη λαθών. Δεν είναι μόνο 100% ε, τα σφάλματα, είναι κάποιε πρημοδοτήσει συγκεκριμένων επιχειρήσεων που είναι ασύμβατε και σε τέτοιε περιπτώσει ζητούμε ανάκτηση των ποσών από του δικαιούχου ή τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τι πέντε χώρε που εντοπίζονται, που δεν έχουν εκπληρώσει το κριτήριο της εξάντε ερεσιμότητας ή όλες τις προϋποθέσεις της εξάντε ερεσιμότητας. Όπως ε, είπα, έχουμε διάφορα σχέδια δράση για την εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Και για αυτές τις ε, πέντε χώρες υπάρχουν ε, ήδη σχέδια δράσης. Μάλιστα, μερικέ δράσει είχαν ήδη εφαρμοστεί στις, κατά την υπογραφή των συμφωνιών εταιρική σχέση και όλες οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες. Επαναλαμβάνω, έχουμε για κάθε χώρα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Παρακολουθούμε την πορεία εφαρμογής αυτών των δράσεων και συμφωνώ πλήρως με τη σύσταση του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε όμως ε, τις πληροφορίες τον Ιούνιο του 2017 για την, το στάδιο ε, εκπλήρωσης των της εξάντερες ημότητας ε, σε αυτά τα σχέδια δράσης και σε, σε περιπτώσεις, στις περιπτώσεις που δεν ε, ισχύουν οι προϋποθέσεις της εξάντε κατά τη στιγμή της ενημέρωσης πρόκειται να προτείνουμε και αναστολή, να επιβάλλουμε αναστολή των μέτρων. Δεν ακούσαμε όμως ποια ήταν τα ενεχόμενα κράτη-μέλη. Ποια είναι. Uh, Νομίζω ότι αναφέροντα το πρόγραμμα δράσεω επιτροπή ε, και το δικαστήριο. Και θα ήθελα να το Ελεκτικό συνέδριο και επί ευκαιρία. Θα ήθελα να ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο που έκανε τόση διαφήμιση στο πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω άλλωστε είχε κάνει και στο παρελθόν για τι δημόσιες προμήθειε. Η Ιταλία, η Ρουμανία, η Τσεχία, η Κροατία και η Σλοβακία από ό,τι γνωρίζω είναι οι πέντε εμπλεκόμενες χώρες. Η Τσεχική Δημοκρατία έχει δώσει ήδη απαντήσεις το 2016 για την πλήρωση όλων των δράσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα δράσης. Για τα άλλα τέσσερα κράτη δεν έχω ακόμη πλήρη ενημέρωση, αλλά θα τα περιλάβουμε στη γραπτή μας απάντηση. Η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό θα προσθέσει κάτι. Κάποιος άλλος, όχι. Ο κύριος Αλή για να ολοκληρώσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, το ελεγκτικό συνέδριο και την Επιτροπή, αλλά και τους αδέλφους. που επισημαίνουν ένα πολύ σημαντικό θέμα, το συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, αλλά και μεταξύ των διαφορών υπηρεσιών της Επιτροπής. Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα έχει μεγάλη σημασία. Περιμένω βέβαια να δω και τις προτάσεις των συναδέλφων που θα ενσωματωθούν στο τελικό έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήσαμε το θέμα αυτό. Τη σημερινή του σημείου αυτό τη ημερική διάταξη. Ε, παρακαλώ να διαβαστούν και οι ευχαριστίε μα ε, για τη ε, συνεργασία και τι απαντήσει. Τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστασία του έναντι των κρατικών ενισχύσεων έχουν τεράστια σημασία. Δυστυχώ, δυστυχώς που βλέπω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Εξατλήσαμε λοιπόν το σημείο 8 και επιστρέφουμε στο 7 της ημερήσιας διάταξης. Έλεγχος του προϋπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μάρκους Πίπερ είναι εισηγητής, έκθεση πρωτοβουλίας και θα λάβει το λόγο για να μας την παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. και για την ευελιξία που επιδείξατε ε, στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θελήσαμε να εξετάσουμε κατά πόσο μη κυβερνητικέ οργανώσεις χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τι τα κάνουν ακριβώς τα χρήματα αυτά που λαμβάνουν. Θα πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι είναι σχεδόν ανέφικτο και αδύνατο να βρει κανείς αξιόπιστα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της το πιστώνω αυτό, κάνει πάρα πολλά για να βρει τα στοιχεία αυτά και να μας τα δώσει, αλλά σας παρακαλώ, δώστε μας τα ονόματα των 50 μεγαλύτερων ΜΚΟ που δεν υποχρεούνται να ε, προβαίνουν σε μία δήλωση διαφάνεια σχετικά με τον τελικό δικαιούχο. Ε, ωραία έκφραση αυτή που έχουμε στα διορθωτικά ταμεία και στα γεωργικά ταμεία. Θέλαμε να έχουμε τους 50 μεγαλύτερους και αυτό δεν κατέστη δυνατό. Είναι ένα από τα πρώτα αποτελέσματα της παρούσης εκθέσεως αυτό. Έχουμε μεγάλα προβλήματα για να βρούμε ε, αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία και για να βοηθηθούμε αναθέσαμε εμεί μια μελέτη σε δευτερογενείς πηγές, όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντίστοιχα έχουμε και τα αποτελέσματα να συνοψίζονται στην έκθεση. Τι συμβαίνει λοιπόν. Είναι μεγάλο το ποσό. Έχουμε ένα στοιχείο από το 2010, που θα ισχύει 1,5 ε, δισεκατομμύριο ευρώ περίπου είναι η χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προπλογισμό. 70% ε, μόλις σε 273 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι κάπως ανησυχητικό. 1,5 εκατομμύριο ε, για κάθε μη αυτή είναι η τάξη μεγέθους σίγουρα θα υπάρχουν πολλές χιλιάδες μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Ευρώπη, λίγες όμως είναι εκείνες που απολαμβάνουν ε, οικονομικής ε, στήριξης ε, αξιόλογο έτσι, βαθμό και ποσά μη ευκαταφρόνητα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τη διαθεσιμότητά τους, κάποιες γενικές παρατηρήσεις τώρα για την ίδια την έκθεση. Θεωρούμε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και στι Βρυξέλλε είναι πολύτιμη βοήθεια για την λήψη πολιτικών αποφάσεων, γιατί πολύ συχνά μας παρέχουν πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις βρούμε από άλλες πηγές. Και θεωρούμε ότι όντως πέρα από την ιδιωτική χρηματοδότηση χρειάζονται και δημόσια οικονομική στήριξη μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έρχομαι τώρα μέσα στα προβλήματα, διότι αναφέρονται και αυτά στην έκθεση και καταλήξαμε στο ευρήμα ότι δεν είναι απρόσκοπτη ε, ε, ε, διαχείριση των κονδυλίων και δεν στοιχειοθετούνται τα πάντα χωρίς προβλήματα και χωρίς κενά. Έχουμε σαν ψηφιδωτό και λείπουν κάποιες ψηφίδες για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Αυτό είναι το πρώτο σημείο κριτικής. Ένα δεύτερο όλο και περισσότερο έχουμε την εντύπωση ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πληρώνονται για ένα συγκεκριμένο έργο, ενώ ε, δουλεύουν με ε, ψευδή στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβολίες ε, διασποράς εσκεμμένης ψευδών ειδήσεων και στη συνέχεια ε, αυτές οι ΜΚΟ ε, χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτά είναι απαράδεκτα. Ναι, ε, και ένα άλλο πρόβλημα και ουσιαστικό και βασικό είναι το γεγονό ότι από ό,τι φαίνεται από την εκτελεστική εξουσία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, υποστηρίζονται ορισμένε μη κυβερνητικέ οργανώσει ή τουλάχιστον λαμβάνουν προσφορά για το πώς να ε, ασκούν πίεση λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους εκπαιδεύουν κιόλας. Ε, υπάρχουν ε, συμφωνίες για στόχους που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ΜΚΟ και ως δημοκράτης ρωτώ με. Επιτρέπονται τέτοια πράγματα να εκπαιδεύει ομάδες λόμπι εκτελεστική εξουσία για να ασκούν πίεση στην νομοθετική εξουσία που είμαστε εμείς. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να το χωνεύσω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τώρα εγώ συνταγματολόγος δεν είμαι ούτε τίποτα τέτοιο, αλλά θέλω να θέσω αυτό το ερώτημα. Αυτό συνάδει με τις ευρωπαϊκές ε, αξίες και αρχές. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι δεν είναι τόσο προβληματικό όσο το αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά χρειάζεται εξέταση. Κάποιες συγκεκριμένες τώρα προτάσεις και αιτήματα για τη διαφάνεια. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία ε, και σαφής ταξινόμηση και ε, κατάταξη των ΜΚΟ. Κάθε γενική διεύθυνση έχει το δικό της σύστημα, πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ ε, την σύγκριση και τον έλεγχο από το να υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα καταχώρησης και ταξινόμησης. Έχουμε κάποιες προτάσεις κάνει για να αυξηθεί η διαφάνεια για το τι θα μπορούσε να αλλάξει και μεταξύ άλλων προτείνουμε Εμεί και στο βαθμό που χρηματοδοτούνται σε ύψος μεγαλύτερο του 10% να το δηλώνουν στους ισολογισμούς τους, στην ιστοσελίδα τους και στο λογότυπό τους να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια ε, από μόνες τους. Ας πούμε, ε, σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ των ε, ηγετικών τους στελεχών, γιατί καμιά φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με εκπλήξεις. Και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει κάπως να δημοσιεύονται και να ε, εντοπίζονται και οι πολιτικές επαφές και η δραστηριότητα λόμπι που ασκούν αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και επίση ενδεχομένω θα μπορούσε να υπάρχει ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό σήμα, μια σφραγίδα ε, για ΜΚΟ που ανταποκρίνονται σε κάποιες ε, προϋποθέσεις και δεσμεύονται και είναι και πιο χαλαρή, πιο εύκολη έλεγχη σε αυτή την περίπτωση. υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται πάντο που είναι η ε, online εγγραφή ενός πιθανού δικαιούχου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να διευρυνθεί. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε και πού ε, καταλήγουν αυτά τα χρήματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες εγκάρσεις, ιδέσεις και πλοκάμια σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μια συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά ε, τα χρήματα αυτά ε, διαχέονται προς μικρότερες μήκυο και θα πρέπει αυτά να τα γνωρίζουμε, πού καταλήγουν και εδώ να υπάρχει ίδια διαφάνεια όπως και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε προτείνει να υπάρχει ένα νέο σύστημα ε, ελέγχου ε, με νέα κριτήρια να μην μπορεί η Γενική Διεύθυνση να κάνει ό,τι θέλει ε, και μέχρι τη διαφάνεια που θα φτάνει στον τελικό δικαιούχο. Δηλαδή ότι στο συγκεκριμένο έργο έφτασαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ίδιο ισχύει και για τα διορθωτικά ταμεία. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία των κρατών μελών και μόνο έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί να τα διεκπαιρεώσει αυτά. Ένα τελευταίο, χωρίς να είναι αυτό λιγότερο σημαντικό, συμπερίληψη εξωτερικών οργανισμών. Δυστυχώ το ελεκτικό συνέδριο μέχρι τώρα δεν έχει ασχοληθεί εντατικά με αυτή την υπόθεση και αυτό μας λυπεί και καλούμε το ελεγκτικό συνέδριο να καταρτήσει ειδική ε, έκθεση ε, για να ασχοληθεί με όλα τα θέματα που, διαπραγματεύεται, που πραγματεύεται συγγνώμη, έκθεση. Ούτε η Όλαφ μας έχει δώσει πληροφορίες για τις ΜΚΟ. Εδώ χρειάζεται καλύτερη πρόσβαση της Όλαφ σε όλα αυτά. Και πάλι, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει επιτελούν σημαντικότατο έργο και πολύτιμο, ιδιαίτερα για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, διότι όταν κανείς επιχειρηματολογεί με διαφάνεια και με πραγματικά ε, γεγονότα και περιστατικά και όχι με ε, αναλήθειε ή ψευδείς ειδήσει, τότε μόνο θα προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σάνεφος Μπάρτ ε, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, συμφωνώ εξ ονόματος ε, συναδέλφου από την ομάδα μου που κολλείται σήμερα και αποσιάζει, αλλά τα έχουμε συζητήσει. Κάναμε ακρόαση, αν θυμάστε, ε, με μεγάλη προσέλευση και ε, το δικό μου συμπέρασμα από την ακρόαση αυτή ήταν ότι όλοι οι παρόντες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρούσαν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τη, τα, της ΜΚΟ. Και λυπάμαι λίγο για την προσέγγιση του συναδελφού Πίπερ, με τον οποίο γενικά συμφωνώ είναι ότι τα βλέπει όλα τόσο μελανά ε, και θέματα που άπτονται τον ΜΚΟ. Έτσι τα, τα περιγράφει με σκούρα χρώματα. Ε, από την άλλη λέει ότι επιτελούν πολύ καλό έργο, πολύτιμο και πάρα πολύ ε, θετικό και το τόνισε και δύο φορές ότι είναι τεράστια σημασία τους, ότι λειτουργούν καλά, ότι έχουν ένα ρόλο για την κοινωνία. Όλα αυτά καλά, αλλά στην έκθεσή του έχει μάλλον ένα αρνητικό τόνο και μια αρνητική προσέγγιση. Και αγαπητέ συνάδελφε Πίπερ, στην έκθεσή σας μιλάτε και με ασέβεια για τις ΣΜΚΙΟ. Διαβάζοντας την έκθεσή σας κανεί, αποκομίζει την εντύπωση ότι έχουν προβλήματα στη λειτουργία τους, πολύ ειδικά, χωρίς να δίνετε τις αντίστοιχες αποδείξεις για όλα αυτά που ισχυρίζεστε. Δεν το βρήκα αυτό στο κείμενο ε, της έκθεσής σας, ούτε στην ακρόαση που είχαμε κάνει εδώ, με πάρα πολλούς ε, συμμετέχοντες που δίρκησε και δύο ώρες μάλιστα. Όταν συζητούμε για μη κυβερνητικέ οργανώσεις, βεβαίως έχει σημασία η διαφάνεια, ε, βεβαίως έχει σημασία ο ανοιχτό χαρακτήρας τη λειτουργία, το αναγνώρισαν και οι ίδιοι σε ΜΚΟ, αλλά υπάρχει αρχή της μη διάκριση. Δηλαδή θα τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από ό,τι άλλους ενεχομένους εκεί και συμμετέχοντες. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτά που λέτε θα ε, επιδεινώσουν τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά το διοικητικό άχθος. Καλό είναι που κάνετε κάποιες συστάσεις Ε, για να ε, αφαιρεθούν τα σφάλματα στη διαχείριση ε, και στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και των κρατικών κονδυλίων και να ξέρουμε και τους τελικούς δικαιούχους, όλα αυτά καλά. Αλλά είναι κάποιες παράγραφοι που παραμένουν ασαφείς. Ας πούμε, στην παράγραφο 6 είναι πάρα πολύ αμφίσιμα αυτά που λέτε. Ε, παραθέτετε κάποιες ε, παραδοχές και σας ερωτώ ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που σας οδηγούν σε αυτή την άποψη ότι δρούν με αυτόν τον τρόπο η ΜΚΟ. Στην παράγραφο 7 απευθύνεστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ειλικρινά τουλάχιστον να μου εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείτε γιατί δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. λογοδοσία, ε, διαφάνεια, ανάληψη ευθύνης, όλα αυτά είναι καλά και ε, ευπρόσδεκτα. Και είμαστε στο πλευρό σας και η ομάδα μου και εγώ, στην παράγραφο 12. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο στιγματίζονται οι ΜΚΟ σε σχέση με άλλες οργανώσεις ως προς αυτό. Στην παράγραφο 12 λέτε ότι υπάρχει δικό πρόβλημα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις όταν πρόκειται για τη λογοδοσία τους. Το ίδιο ισχύει και για την παράγραφο 25. Μα τα περισσότερα χρήματα που παίρνουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι πόροι που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση κάποιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ συχνά πρόκειται για θέματα και έργα αναπτυξιακής συνεργασίας. Άρα ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων αυτών δεν ε, τον δαπανούν για να επηρεάσουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν τέτοιες ε, ΜΚΟ και εκεί υπάρχει το Μητρό Διαφάνειας, αλλά για χρήματα τα οποία δαπανούν επί τόπου οι ίδιες οι ΜΚΟ με τρόπο πάρα πολύ αξιοπρεπή και αξιόλογο στην αναπτυξιακή βοήθεια, ε, δεν χρειάζεται αυτό το ίδιο Μητρό Διαφάνειας. Στην παράγραφο 34, σε ό,τι αφορά και εμένα και την ομάδα μου, πρέπει να σας πω ότι είναι τελείως απαράδεκτη. Γιατί εκεί γράφεται ε, ρητά ότι υπάρχ, υπάρχει απάτη στη διαχείριση, χωρίς να φαίνεται στοιχεία αποδεικτικά. Τέτοιες παράγραφοι πραγματικά είναι αρνητικές για την έκθεση και δεν καταλαβαίνω πού το βασίζεται αυτό για να το ισχυρίζεστε. Το βασικό πρόβλημα ποιο είναι κύριε Πίπερ και σας ερωτώ και φάνηκε και από την ακρόαση. Είναι ο ορισμός ο ίδιος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όταν μιλάτε στην έκθεσή σας για ΜΚΟ, τι ακριβώς εννοείτε. Γιατί στην ε, ακρόαση ήταν ακαθόδες αυτό το θέμα και το παραδέχομαι. Υπάρχει ζήτημα με τον ορισμό. Εσείς λοιπόν όταν μιλάτε για μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σε τι αναφέρεστε, σε επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις ε, εκπροσώπων Business Europe, ας πούμε, επαγγελματικών κλάδων. Μιλάτε για ιδρύματα, για Ινστιτούτα, για οργανώσεις, που, ομάδες πίεσης που επηρεάζουν ή θέλετε να κατονομάσετε ποιες ΜΚΟ είναι αυτές ή υπάρχουν κάποιες άλλες που είναι μη κερδοσκοπικές, υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που είναι ε, πάροχοι υπηρεσιών και κάποιοι άλλοι που ε, απλώς ε, θέλουν να προωθήσουν ένα ζήτημα που είναι παροχή συμβουλών ή λεγόμενες advocacy. Ε, αυτά ρωτώ για να μπει στη σωστή τροχιά η έκθεση και να συνεννοηθούμε όλες οι πολιτικές ομάδες και να πούμε ότι πρόκειται για αυτές τις ΜΚΟ, τις συγκεκριμένες. Αυτές χαρακτηρίζουμε τις συγκεκριμένες οργανώσεις μη κυβερνητικέ και όχι ό,τι να είναι. Ε, στην πρώτη παράγραφο μιλάτε ε, για τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό είναι φλουαρτιστικ. Ε, είναι έτσι μια καλλιτεχνική θολούρα γενική που θολώνει την έκθεσή σας και της αφαιρεί και ισορροπία. Σίγουρα θα κάνουμε τροπολογίες και οπωσδήποτε θα, θα το δούμε και διμερώς για να διασκεδάσουμε οποιασδήποτε παρεξηγήσεις ενδεχομένω έχουν ε, δημιουργηθεί. Και ο συνάδελφο Πυρίσκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πόχετο που είναι ο σκιώδης ηγητής. Ο κύριος Πόχε που είναι ο σκιώδης ηγητής μου ζήτησε μια και απουσιάζει να παρουσιάσω τις απόψεις του. Καταρχήν αναγνωρίζει την αξιόλογη σχέδια, το, το αξιόλογο σχέδιο έκθεση, την αξιόλογη έκθεση και παρόλα αυτά έχει μερικές ε, ανησυχίες ε, και κάποιες επικρίσεις τις οποίες και θα υποβάλει με τη μορφή τροπολογιών προκειμένου να διορθώσει κάποια σημεία που κατά τη γνώμη του είναι συζητήσιμα. Καταρχήν θεωρεί ότι η έκθεση θα πρέπει να εδράζεται σε αδιάσυστα και αντικειμενικά στοιχεία και φαίνεται ότι πολλές από τις πηγές που αναφέρονται στην έκθεση είναι αμφισβητήσιμες ως προς την αμεροληψία τους παρόλο που στι αιτιολογικές σκέψει παρέχονται κάποια στατιστικά στοιχεία για τα οποία θα ήθελα διευκρινήσεις ο κύριος Πόχε και να μα πει ο εισηγητή ε, τι πηγέ του. Δεύτερο σχόλιο για το σχέδιο έκθεσης αφορά την αρχή της αναλογικότητας. Η έκθεση ε, υποβάλλει πλειάδα απαιτήσεων προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Μερικέ είναι ουτοπικέ, εξαιρετικά επαχθεί και δυσανάλογε ω προ τον κίνδυνο που εντοπίζει ο εισηγητή. Αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε το σύστημα και όχι να το ε, επιβαρύνουμε με περαιτέρω διατυπώσει ώστε να το κάνουμε αναποτελεσματικό, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένου τομεί όπου είναι δυνατέ και απαραίτητε οι βελτιώσει δεν θα πρέπει να παρεξηγείται εδώ το σκιώδη εισηγητή, γιατί θεωρεί ότι μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι και να δικήσουμε κάποιες ε, αξιώσεις, αρκεί αυτές ε, να είναι προσγειωμένες και ρεαλιστικές, γιατί η προσθήκη νέων φραγμών θα παρεμποδίσει την άσκηση του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις αδυναμίες που έχει το σύστημα και όχι σε συγκεκριμένες μη κυβερνητικέ οργανώσει. Γιατί το συγκεκριμένο σύστημα χορήγηση επιδοτήσεων παρά είναι επαχθέ, ιδιαίτερα για τι μικρέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και έχουμε και. Ο σκιώδη ηγετή έχει κάποια προβλήματα με συγκεκριμένε παραγράφου. Καταρχήν την παράγραφο 5 και την ανακατανομή των κονδυλίων εντό συγκεκριμένων ενώσεων. Ο σκιώδη πιστεύει ότι σε πολλέ περιπτώσει είναι λογικό για την ε, ε, ε, κεντρική μη κυβερνητική οργάνωση να μοιράσει τα κονδύλια προς τις ε, θηγατρικές κατά κάποιο τρόπο, εφόσον όμως στηρούνται οι έλεγχοι απαραίτητη και επιτρέπεται τέτοιου είδους ε, υπεργολαβία. Επίσης, η δικτύωση είναι υποφελής και για τις οργανώσεις αυτές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εξασφαλίζει καλύτερη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Για την παράγραφο 6 ακούσαμε ήδη κάποια σχόλια ο κύριος Πόε θα ήθελα να επισημάνει ότι είναι ασαφές ε, τι προτείνει ο εισηγητής. Να ισχύσει παράγραφος 6 μόνο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή για όλους τους δικαιούχους των κυρωτικών κονδύλιων. Γιατί αν ισχύει το πρώτο, εμ, απο, αποβαίνει βάρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αν συνιστά διάκριση και αν το επεκτείνει σε όλου του δικαιούχου, είναι υπερβολικά επαχθέ το μέτρο που προτείνει. Επίσης, μερικές φορές οι φιλοδοξίες παρά είναι υπερβολικές. Στο σημείο 7 αναφέρονται κάποιες συγκεκριμένες μορφές βάρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζονται σε αμφισβητήσιμες πηγές και θα θέλαμε διευκρινήσεις για το πόσο ευθέτη είναι τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το, το τμήμα για τη διαφάνεια, ο, ο ε, είναι υπέρ ενός ε, μητρώου ε, πιο ρωμαλαίο μητρό ε, διαφάνεια. και επίση, η καταχώρηση στο μητρό αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για, όλες, για όλους τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων. Και επίση θα πρέπει ε, να γίνεται τακτικός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, το θέμα της, διαφα... της διαφήμισης ε, το... της σχετικής υποστήριξης θα πρέπει να... να εξασφαλίζεται από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και εδώ θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις για την πρόταση του συγητού σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας ε, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε κάτι τέτοιο να εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των δικαιούχων και όχι μόνο στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ίδιο ισχύει και για το τμήμα που αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Και φυσικά και εκεί συμφωνούμε με την ανάγκη βελτιώσεων, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιβάλλεται τόσο περιττό άχθος προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα, σοβαρό κατά τη γνώμη του και του στοιχείου ε, ε, ε, είναι οι ασυνέπειες μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι επιμέρους δι... γενικές διευθύνσεις χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες, κάτι τέτοιο αποβαίνει εις βάρος της διαφάνειας. Θέλουμε εναρμονισμένους κανόνες για τα κοινοτικά κονδύλια. Επίσης θα πρέπει να προσφέρεται εκπαίδευση προς τις ευρωπαϊκές ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις για να ενημερωθούν καλύτερα για τους κανόνες και θα θέλαμε να μας διευκρινίσει ο εισηγητής που ε, ε, αν στην παράγραφο 8 είναι υπέρ της ε, κατάρτισης ε, σε θέματα δημοσιονομικού κανονισμού, γιατί αν αυτό προτείνει, ίσως καλό θα ήταν να διατυπώσουμε την παράγραφο 8 για να διευκρινιστεί αυτός ο σκοπός. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα προβληματισμού του σκιώδου συγγητού. Σας ευχαριστούμε κύριε Πυρίνσκι. Θα ήθελα να αντικαταστήσω... Την πρόεδρο για λίγο, αλλά θέλω και εγώ να λάβω το λόγο. Τρεις ερωτήσεις. Δεν μπόρεσα να λάβω μέρο στο εργαστήριο που είχατε οργανώσει. Δυστυχώ φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσο μιλούσατε, γεννήθηκαν στο μυαλό μου κάποιε απορίε. Αντίστοιχε με αυτά που επισήμανε και ο Μπάρτ σε παραδείγματι, είπε ήταν πολύ δύσκολη συλλογή πληροφοριών. Τι πηγέ χρησιμοποίησατε, δημόσια προσβάσιμες πηγές, ε, τι στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, και τι πηγές αξιοποιήσατε για το σχέδιο. Δεύτερον, όπως είπε ο κύριος Στάς, πώς ορίζονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην Ευρώπη επιμένουμε ιδιαίτερα, όπως είπατε και εσείς, ε, για το, για το μητρό των λόμπι των ομάδων πιέσεως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καλύπτονται όλες οι κυβερνητικές οργανώσεις, και όλες οι κυβερνητικές οργανώσεις είναι ομάδες ε, πιέσεως. Υπάρχουν ε, ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν και ε, εμπορικά συμφέροντα μέσα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Παρακαλώ λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς κάνετε αυτό πώς, ε, ποιον ορισμό ακολουθείτε και πώς κάνετε τη διάκριση του ποιος, έχει, ποιος είναι η κυβερνητική οργάνωση και ποιος όχι. Μια και αναφέρατε επίση στην Όλαφ στην εκθεσή σας. Ε, υπάρχουν κάποιες ενεξελίξει έρευνες της Όλαφ εις βάρος μη κυβερνητικών οργανώσεων ή έχετε κάποιες πληροφορίες για τέτοιου είδους ε, έρευνες από το παρελθόν εις βάρος μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Σε μεγάλο βαθμό εστερνίζομαι την ανάλυση του κυρίου Πίπερ. Δεν τον ξαφνιάζω φαντάζομαι. Στο σημείο 1 ιδιαίτερα ο εισηγητής ε, επισημαίνει τη σημασία που έχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει για την εκτέλεση των κοινωτικών πολιτικών. Και συμμερίζομαι απόλυτα αυτό το στόχο και αυτή την δήλωση που κάνει ο κύριο Πίπερ. Και μάλιστα έλαβα μέρο στη συζήτηση για την χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και άκουσα τις ανησυχίες και τον προβληματισμό τους. Επίσης, είναι σημαντικό το ποσό που αναφέρουμε το 1,5 δισεκατομμύριο δηλαδή ευρώ, που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον κύριο Στάες ότι ε, η δική μας, η δική μας επιτροπή πρόσφατα ανέκρινε την έκθεση Young. Ε, Είχαμε και την έκθεση Σέλερ, την οποία επίσης εγκρίναμε. Και συμφωνώ να μην ε, ε, μεταχειριζόμαστε αρνητικά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να μην θεσπίζουμε διακρίσεις βάρος τους. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί μόλις συζητήσαμε την έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και ζητούμε εξηγήσει από τα κράτη-μέλη. Γιατί όχι και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Με προβλημάτισε κάπως και με, με, θορύβησε αυτό που είπατε, ότι είναι αδύνατο να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των σημαντικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό πραγματικά με ανησύχησε ιδιαίτερα. Και επίσης είπατε ότι η πολιτική αυτή είναι συνεπής και σχετικά συνάρτη. Εγώ θα ήθελα τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στην πολιτική αυτή και να έχουμε πολιτικές ελέγχου και παρακολούθησης. Και επευκαιρία για να μην μακρηγορήσω, γιατί φαντάζομαι ότι ο εισηγητής θα απαντήσει στις απορίες μας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να απαντηθεί μία ερώτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ναι, και μιλούμε για την ανάγκη πιο ακριβώς στοιχείων. Τι έλεγχοι γίνονται για τη χρηματοδότηση αυτή το, αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπήρξαν παρατυπίες, γιατί προηγουμένως ρωτήσαμε τι έγινε με τα 137 δισεκατομμύρια ε, κρατικών ενισχύσεων ε, δυνάμει της ε, πολιτικής συνοχής. Τι έγινε με αυτό το 1,5 δις για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις διατυπώθηκαν, παρά τι έγινε, ανάκτηση κάποιων ποσών και τι μηχανισμούς ελέγχου χρησιμοποίησατε τα τελευταία χρόνια για να έχουμε μια ιδέα της τάξης μεγέθους των ποσών που συζητούμε. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι η έκθεση Πίπερ πραγματικά θέτει το δάκτυλο επί του τύπου των ήλων. ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Και γι' αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε στοιχεία στη διάθεσή μας. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με την ανησυχία του εισηγητού ότι είναι δύσκολο να αποκτήσουμε αξιόπιστα στοιχεία για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ που όπως ε, είπε και ο συγητής, συμφωνώ μαζί του, είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι σημαντικός παράγοντας και συντελεστής ε, στην εκτέλεση αυτών των πολιτικών, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε την συνέπεια, τη συνοχή μεταξύ της χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων και των αρχών μας, γιατί θα ήταν εξωφρενικό μέσω μηχανισμών ανεξέλεγκτων να χρηματοδοτούμε πολιτικές και στόχους που δεν συνάδουν με τους στόχους της συνθήκης. Να μην σας επιθυμίσω τι φάση βρίσκεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πραγματικά θα ήταν εξωφρονικό και παράλογο να χρηματοδοτούμε δραστηριότητες μέσω μηχανισμών που διεφεύγουν το ελέγχου μας, να χρηματοδοτούμε σκοπούς που αντιβαίνουν στις αξίες της συνθήκης. Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, κύριε Κελκασάδο, Κομισιόν. Α, κύριε Αλή, με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Ναι, ο κύριος Τάκουλας και ο δεσηγητής μου ζήτησε να αναλάβω το λόγο εκ μέρους του. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ο σκιώδης κύριος Τάκουλα θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία όταν συζητούμε για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών οργανώσεων ε, ε, ζώμη όχι μόνο στα κριτήρια της διανομής ε, των χρημάτων, αλλά και τη... το σκοπό για τον οποίο διατίθεται τα χρήματα αυτά και ο κ. Στάκουλα λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να απορρίπτει χρηματοδότηση σε περίπτωση που οι στόχοι της μη κυβερνητική οργανώσεως στρέφονται κατά των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω, η ευθύνη για την παρακολούθηση τη τρίση των στόχων αυτών θα πρέπει να είναι δεδομένη και η χρηματοδότηση και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάγεται σε αυτού του όρου. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι όταν συζητούμε για τη χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει ε, εν γέννη να αποφεύγεται ο γραφειοκρατικό ε, φόρτο. Δεν πρέπει οι μικρέ δηλαδή μη κυβερνητικέ οργανώσει να επιβαρύνονται δυσανάλογα. Οι μικρότερε οργανώσει επίση πρέπει να συνυπολογίζονται και κατά την ε, χάραξη των νέων κανόνων για τη διαφάνεια, καθώς είναι εκείνες οι οποίες ε, περισσότερο ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία. Ο κύριος Στάκουλας σημειώνει επίσης ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι τα ίδια για όλες τις οργανώσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Χιλχασάδο. Ευχαριστώ. εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα ήθελα να σημειώσω ότι η έκθεση αλλά και όλα τα θέματα που συζητούμε και που συζητήσαμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο η ανταλλαγή ε, θέσεων, η επικοινωνία με τον εισηγητή, όλες οι επαφές μας είχαν ένα στόχο, τη συλλογή των στοιχείων, των πληροφοριών και συμφωνούμε μαζί σας ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν ουσιώδη ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να είναι μοναδικοί βέβαια παράγοντες. Οι φορεί υλοποίηση έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό τείνουμε να συμφωνούμε με ορισμένα από τα σχόλια που εκφράστηκαν σήμερα εδώ. Έχουμε την εντύπωση ότι η έκθεση έχει μια αρνητική χρειά ως προς τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. στη διευκόλυνση της υλοποίησης της πολιτικής ε, των θεσμικών οργάνων. Με έκπληξη μάλιστα διαπιστώνουμε ότι κάποιες από τις συστάσεις του εισηγητή που αφορούν μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι σε μεγάλο βαθμό πολύ καλές βεβαίως ε, και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις ε, λάβει υπόψη, να τις ενισχύσει, να τις εμπλουτίνει προκειμένου να ενισχύσει την ε, διαφάνεια. Λαμβάνουμε σοβαρά μέτρα. Το σύστημα χρηματοοικονομικής διαφάνειας FTS που έχει υιοθετηθεί από το 2010 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βελτιώνεται βήμα το βήμα, έχει ακόμα βέβαια περιθώρια βελτίωσης. Επιτρέψτε μου ωστόσο να αναφερθώ σε κάποια σημεία και της έκθεσης ε, στο, στη γράψη στο γραπτό κείμενο, αλλά και κάποιον από τους εδώ παρισταμένους βουλευτές. Ε, θέματα λογοδοσίας και ελέγχου, επί παραδείγματι, το δράση των κυβερνητικών οργανώσεων, που είναι και αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου σας. Αναφέρθηκε ότι είναι εμπλεκόμενοι φορείς οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά ίσονες εμπλεκόμενοι φορείς από τις πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με την ε, εκτέλεση των προγραμμάτων από μια κυβερνητικέ οργανώση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει αυτή η κατηγορία εμπλεκόμενων φορέων να τύχει διαφορετική μεταχείριση από ό,τι άλλοι εμπλεκόμενοι φορεί. Θα λάβει βεβαίω υπόψη κάποιε από τι συστάσει τη εκθέσεω προ πιο αυστηρή μεταχείριση σε σχέση με άλλου. Λαμβάνεται υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει ένα πλήρες σε σύστημα ελέγχων στηριζόμενο στην ανάλυση κινδύνου με ε, τη χρήση μια σειράς εργαλείων είτε για αντίδραση είτε για αξιολόγηση ε, παρατυπιών, απατών ε, ή προβλημάτων άλλων και βέβαια έχει στη θέση της και μέτρα αποκατάστασης και Άλλου τρόπους δράσης έναντι μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και κάθε άλλου φορέα, περισσότερο προς τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και κάποιε από τις προτάσεις που έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ έντονες δυσκολίες για τους εμπλεκομένους φορείς. Παραδείγματι, η διάθεση εκθέσεων για το προσωπικό, η ανάλυση του δικτύου. Ναι, συμφωνούμε ότι μερικές φορές πρέπει, χρειάζονται την ανάπτυξη δικτύων οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά πρέπει πάντα να είναι ορατό και, ε, ορατός και ο στόχος για τον οποίο ε, εργάζονται και για τον οποίο θα λάβουν τη σχετική χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται δηλαδή να δεχθούμε να καταβάλουμε οδήποτε ποσό σε υπεργολαβίε, όπω είπατε εσεί, ή κάτι άλλο, εάν προηγουμένω δεν έχει κοινοποιηθεί και εγκριθεί ο, ο στόχο που εξυπηρετεί η μη κυβερνητική οργάνωση. Άλλωστε, αυτό είναι κομμάτι τη εκ των προτέρων διαφάνεια, όταν ε, δηλαδή δημοσιεύεται ε, το πεδίο δράση και ο στόχο. Ο σκοπός. Επίσης, η Επιτροπή Ιδιαίτερα στην πρόταση αυτή για τον νοσομικό κανονισμό που προσπαθούμε να εισαγάγουμε, ε, προσπαθεί και να λάβει υπόψη τη διάσταση του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της διευκόλυνσης των διαδικασιών και πιστεύουμε ότι ορισμένες από τις συστάσεις της εκθέσεως δεν βαίνουν προς τον ίδιο στόχο. Σημαντικό επίσης ε, είναι το εξής, η εναρμόνιση των κανόνων και η κεντρική οργάνωση του συστήματος διαχείρισης. Έχετε δίκιο βεβαίω. Χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση. Συγκεκριμένα προγράμματα μπορεί να παρουσιάζουν αποκλήσει μεταξύ του. Και έτσι μπορεί οι εμπλεκόμενοι φορεί, εκείνοι δηλαδή που εργάζονται σε διαφορετικά προγράμματα, να βρίσκονται σε μηχανία, να μην βλέπουν τι διαφορέ κτλ. Και βέβαια αναλόγω να μην αντιλαμβάνονται και ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κανόνε. Ο δημοσιονομικό όμω κανονισμό προβλέπει και ε, περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία, ένα συνεκτικό πλαίσιο και τίνει προ την εναρμόνιση των κανόνων, τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Όπω σε παραδείγματι έχουμε όλου του κανόνε για τι δημοσίευσει εκ των προτέρων, εξάντε, τη ε, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο, τη δημοσίευση των στοιχείων, των υποχρεώσεων για τήρηση βιβλίων, εκθέσεις, όλα αυτά καταγράφονται στο δημοσιονομικό κανονισμό όπως έχει τώρα. Πάλι όμως, περαιτέρω εναρμόνιση και πάντως καλύτερη διαφάνεια θα εξασφαλίσουμε αν προχωρήσουμε προς την ηλεκτρονική κατάθεση και διαχείριση, ηλεκτρονική διαχείριση των χορηγιών αυτών. Έτσι λοιπόν με ένα μοναδικό κατά προτίμηση σημείο επικοινωνίας, ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή εισόδου. Μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών ε, κρατικών προμηθειών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει με κυβερνητικές οργανώσεις. Προσπαθούμε να διευρύνουμε το πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος με την ψηφιοποίηση ασφαλώς θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και, περισσότερα, και καλύτερα στοιχεία και για σας. Και επίσης εν τέλει για την ορατότητα της χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αισθάνεται κατάπληξη για κάποιες από τις εκτιμήσεις τις οποίες προβαίνει η έκθεση, γιατί η ορατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που έχουν λάβει με κυβερνητικές οργανώσεις και βέβαια όλοι οι ε, εμπλεκόμενοι φορείς γενικά, είναι υποχρεωτική. Και άλλωστε η σχετική ενημέρωση υπάρχει ήδη προκαταβολικά στις ε, λεπτομερείς διατάξεις της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέρον, αλλά και μέσα στον κανονισμό. Και στις συμβάσεις διορθώνει ο Μιλήτρια συγκεκριμένα που υπογράφουν οι δικαιούχοι. Ρητά αναφέρεται ότι πρέπει να δημοσιοποιούν το γεγονός ότι έχουν λάβει ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρόκειται για κομμάτι και των όρων ε, λειτουργίας και δράσης μας, αλλά και των ελέγχων μας. Αν αποδειχθεί δηλαδή ότι δεν έχουν γίνει σχετικές δημοσιοποίησεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει και το πράττει μέτρα διορθωτικά. Κάποια μόνο αναφερθήκατε στο θέμα του ορισμού, του τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Μη κυβερνητική οργάνωση είναι βέβαια ένα πάγιο, ένας πάγιος προβληματισμός αυτός. Υπάρχουν και μελέτες, έχουμε και κάποιες προτάσεις. Ε, ενδέχεται όμως αυτό να αποδειχθεί μη, παραγωγικό γιατί το νομικό πλαίσιο, η κατάσταση ε, στα 28 κράτη-μέλη είναι τόσο διαφορετική από το ένα κράτο στο άλλο, που δίνει είναι δυνατόν σήμερα τουλάχιστον στην τρέχουσα εποχή να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μα εξασφαλίσει, θα μα επιτρέψει ενιαίου ορισμού. Άλλωστε δεν στοχεύουμε σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν από μια περίπου πενταετία προσπάθησε μέσα από το σύστημα το λογιστικό που ακολουθούμε να κάνει τη διάκριση μεταξύ των κερδοσκοπικών και μη οργανώσεων. Όπως όμως πολύ εξημών ε, επισημάνατε, ε, οι μη, οι μη κερδοσκοπικές ε, οργανώσεις δεν είναι όλες μη κυβερνητικές. Επομένως προσπαθούμε να βρούμε κάποια άλλη λύση, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή κοινό ορισμό δεν είναι δυνατόν να προκύψει. Και για να επανέλθω στη διαφάνεια και να ολοκληρώσω το σύστημα βεβαίως ε, για τη διαφάνεια του FTS και γενικά η παρουσία υποβολή των δυνατών περισσότερων στοιχείων και δεδομένων ε, βοηθούν ασφαλώς τη διαφάνεια, προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα ακολουθώντας τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζουμε ότι και με την ψηφιοποίηση της διαχείρισης ε, και βέβαια της υλοποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα είμαστε σε θέση στο μέλλον να σας προσφέρουμε πολύ πιο ακριβείς πληροφορίες. Κυρία Τλαβάκοβα, ευχαριστώ. Ο κύριος Πίπερ για να τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Απαντώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. διότι υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις ε, ή και σφάλματα. Δεν ξέρω εσύ και εμένα παρανοείτε την έκθεσή μου. Εγώ πουθενά δεν μιλώ για απάτη. Πουθενά δεν τις κατηγορώ ότι εξαπατούν. Το μόνο που θέλουμε είναι μεγαλύτερη διαφάνεια από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και όταν ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μα είναι υποχρεωμένες να αποδεικνύουν ε, που ε, δαπανούν τα χρήματα αυτά, ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, δεν λέω. Αλλά αυτά συμβαίνουν ε, κρυφά. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως βουλευτές, δεν έχουμε καμία πρόσβαση, δεν μπορούμε να δούμε τι έχετε συμφωνήσει ως προς το στόχο ε, της δαπάνης αυτής και προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι δεν το θεωρεί καθόλου πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάκριση των εξουσιών, εγώ έμαθα στο σχολείο νομοθετική, εκτελεστική, ε, δικαστική εξουσία. Και εδώ ε, είναι προφανές και αυτονόητο λέτε να ε, εκπαιδεύει τα λόμπι η εκτελεστική εξουσία για το πώς μπορούν να βελτιωθούν στις επιδόσεις άσκης πίεσης προς κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Και δεν υδρώνεται αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ χρειάζεται να το κοιτάξουμε αυτό. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε Μάλλον, να το πω αλλιώς. Συμφωνώ με αυτό που είπε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι αυξάνεται ε, το διοικητικό άχθος. Δεν διαφωνώ, αλλά θα πρέπει να ε, υπάρχει ενιαία διαδικασία ε, υποβολή των διαφόρων δικαιολογητικών και παραστατικών για να μπορεί και ένας εξωτερικός παρατηρητής να τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό το αίτημα είναι θεμητό και δικαιολογημένο. Αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα FTS για την οικονομική διαφάνεια. Ας το αξιοποιήσουμε, ας το αναπτύξουμε και ας έχουμε μια ενιαία μορφή ε, λογιστικού ελέγχου που όλοι να ακολουθούν την ίδια ε, οδό και θα έχουμε προχωρήσει προς τους συναδέλφους τώρα για τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν συμφωνώ καθόλου με τα στοιχεία που μας δίνουν. Δεν πήραμε καθόλου στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναθέσαμε μια μελέτη σε εξωτερικούς ε, συνεργάτες που πήγαν και με κόπο ζητούσαν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι δεν πήραν τίποτα. Με εξαίρεση το πρόγραμμα ε, Horizon ε, και τα διαρθρωτικά ταμεία που έχουμε υποχρέωση κοινοποίηση του τελικού δικαιούχου και εκτός από τα γεωργικά ταμεία που ισχύει το ίδιο, υπάρχουν κάτι λίγα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας και περιβαλλοντικά και θέλαμε να έχουμε τον κατάλογο των ε, μεγαλύτερων οργανώσεων που παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Είναι μια απλή ερώτηση. Εμεί τώρα κυνηγάμε την ουρά μας και δεν μας δίνουν τα στοιχεία. Και λέω και προς την κυρία ε, συνάδελφο των Φιλελευθέρων, την κυρία Μαρτίνα ε, Τλαμπαϊόβα, ότι χρειάζεται καλύτερη στάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερη βούληση. Ούτε θέλω να αξιολογούμε και να ελέγχουμε όλους τους ενεχομένους και όλα τα λόμπι, μόνο αυτούς που χρηματοδοτούμε. Δεν είναι δικαιολογημένο αυτό να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να την απαιτούμε κιόλας. και να βλέπουμε ποια είναι η στρατηγική πολιτική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την ελέγχουμε πάρα πολύ αυστηρά. Και όχι κατά το δοκόν. Δηλαδή αυτό που φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκόπιμο, αυτό είναι το κρίσιμο. Και πού είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επειδή τα θεωρεί όλα αυτά σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνούμε κι εμεί. Υπάρχουν λόμπι που δουλεύουν με ψευδείς ειδήσει κατασκευασμένε και είναι γνωστό αυτό, αποδεδειγμένο και στρέφονται και κατά ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και αυτό είναι γεγονός και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Δηλαδή τους αντιπάλους μας τους χρηματοδοτούμε και από πάνω. Ε, θα πρέπει να οξυνθεί λίγο η αίσθηση του προβλήματος και η συνειδητοποίηση του προβλήματος από όλους τους ενδιαφερομένους. Και σε ε, σχέση με τα όσα είπε ο Μπάρτ, σε πολλούς τομείς έχει ε, πραγματικά περιπλακεί το σύστημα πάρα πολύ και είναι υπερβολικές οι ε, ρυθμίσεις και οι απαιτήσει. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου αν θέλεις να τα ξαναδούμε και να τα διορθώσουμε από κοινού στην έκθεση και να τα απλοποιήσουμε ουσιαστικά. Ο συνάδελφος Σαλαφράγκα προς την ίδια κατεύθυνση επιχειρηματολόγησε, ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν, ορισμός των ΜΚΟ Εμένα δεν με νοιάζει ο ορισμός, δεν τον χρειάζομαι. Αλλά να έχουν κάποια κριτήρια ε, σύμφωνα με τα οποία να κρίνονται και να έχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Με χαρά περιμένω τη συζήτηση, τις τροπολογίες και τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε εδώ τη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τώρα αρχίζει η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού για ε, δημοσιονομικό κανονισμό και θα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλες τράπεζες. Εγώ που είμαι συγκήτρια θα μπορούσα να είχα κάνει αυτή τη συζήτηση στο γραφείο μου, αλλά θεώρησα σκόπιμο να τα ακούσουμε όλοι και να γίνει μια κοινή συνεδρίαση. Καλά θα ήταν να εισέλθουν και οι συνάδελφοι.